Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Είναι 9 και 20 πια. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς με μια καλημέρα σε όλους και μετά με την ημερήσια διάταξη στην οποία θα κάνουμε μια μικρή, μικρή τροποποίηση μετά την ώρα των ψηφοφοριών ελπίζοντας ότι θα έχω αρκετό κόσμο στην αίθουσα θα ήθελα να συμπληρώσουμε ένα σημείο πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για ένα περιορισμένο ποσοστό ε, ειδικού φόρου για το ρούμι που κατασκευα... παρασκευάζεται στην Γουαδελούπη Μαρτινίκα Ρεουνιόνο. Αυτό λοιπόν θα το δούμε αμέσως μετά τις ψηφοφορίες. Επίσης υπενθυμίζω ότι έχουμε μετάδοση μέσω του διαδικτύου, της συνεδρίασης, με web streaming και επίσης ότι τα ωράρια που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη είναι μόνο ενδεικτικά. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, προχωρώ στο επόμενο σημείο, την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 7ης Νοεμβρίου, τα έχετε λάβει και ως συνήθως, εάν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις, θα τα θεωρήσουμε εγκεκριμένα στο τέλος συνεδρίασης Και πάμε στο σημείο 3, ανακοινώσει της Προέδρου, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Οι αποφάσεις των συντονιστών, ε, όπως θα προκύψουν σήμερα, θα σας ανακοινωθούν στην προσεχή συνεδρίαση μετά το νέο έτος. Και με αυτά επιτρέψτε μου να περάσω το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης με τον κύριο Ομάρζε, Γιούμου Ομάρζε, βέλτιστη αξιοποίηση των από απόκεντρων περιοχών μέσω τη δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στα διαθροτικά ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μπορεί να μην είμαστε πολύ άριθμοι σήμερα. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να προβούμε σε μια πλούσια και ποιοτική ανταλλαγή απόψεων για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας που αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Καταρχάς επιτρέψατε μου να καλωσορίσω εδώ μια αντιπροσωπεία του Περιφερειακού ε, ε, Συμβουλίου που έχουμε από την Γουαδελούπη ήρθαν να παρακολουθήσουν τις εργασίες μας σήμερα. Η Επιτροπή μας συνηθίζει τακτικά να εκδηλώνει ενδιαφέρον, να εκφράζει το ενδιαφέρον της για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, δεδομένου ότι οτιδήποτε αφορά το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ανήκει στις α, καθήλυνα αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Συχνά, ωστόσο, οι εξόχως απόκεντρες ε, περιφέρειες εξετάζονται υπό το πρίσμα του σεβασμού του άρθρου 349 μόνο, με την δυνατότητα για ε, παρεκκλήσει, εξαιρέσει ή λήψη υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αυτών των περιοχών μα. Είναι άκρο απαραίτητη η προσέγγιση αυτή ασφαλώς, γιατί ακρο απαραιτητη ότι έχουν καθυστέρηση ανάπτυξη αυτές οι εξόχως περιφερειακές ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές και χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους και οι ανάγκες τους. Ωστόσο σήμερα πιστεύω ότι θα πρέπει να ανοίξει μια νέα φάση στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξόχων απόκεντρων περιοχών. Όταν δούμε λοιπόν τα όσα χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξόχως κέντρων περιοχών μέχρι σήμερα είναι μια απόσταση μεταξύ περιφερειακής και γεωργικής πολιτικής. Πιστεύω ότι σήμερα πρέπει πια να ανοίξουμε το φάσμα των στόχων μας, να το διευρύνουμε με νέους στόχους που θα επιτρέψουν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να ενσωματωθούν καταρχάς καλύτερα στην εσωτερική αγορά, αφετέρου δε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που γεννά και η Ευρωπαϊκή και η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη στρατηγική, όπως την άλλωστε την έχουν προδιαγράψει και οι ίδιες οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και με τις ε, εκθέσεις πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκεκριμένα του Νούνο Τεκτσερά και πιστεύω ότι οι φιλοδοξίες μας, αντικείμενο όλος της έκθεσης, θα επιτρέπει μια πρακτική προσέγγιση ώστε όλες οι κοινοτικές ε, πολιτικές να επιτρέψουν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να ε, επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο. Και το δεύτερο, ότι πολύ συχνά έχουμε την αίσθηση ότι η σχέση που συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, μακρινή της περιφέρεια ε, είναι μια ε, σχέση αλληλεγγύης. Αυτό ισχύει όντως, εν μέρη όμως. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εγγράφονται και στο επίκεντρο των στόχων που ε, καταγράφει ως δικούς της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι επενδύσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές αποβαίνουν εις όφελος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί παραδείγματι, στην βιοπικιλότητα δεν είναι δυνατόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους αυτούς χωρίς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, χωρίς τις ε, και τα εδάφη, τα υπερπόντια. Ξέρετε ότι στην ε, συμμετοχή στους στόχους της ε, κλιματικής αλλαγής μπορούν να διδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο οι απόκεντρες ε, περιοχές. Το ίδιο στην προστασία του, ε, των κοραλιογενών υφάλων στην πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές. Το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω. Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα εδάφη και ε, υπερπόντια εδάφη και κτίσεις είναι αυτά τα οποία μπορούν να δώσουν νέα διάσταση και βέβαια νέες δυνατότητες ανάπτυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά είναι τα θέματα στα οποία μπορούμε να δούμε την παρουσία αυτών των εξοχών απόκεντρων περιοχών, εγκαταλείποντας πιστεύω ε, την φαταλιστική αυτή ή την ε, μίζερη προσέγγιση ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ως μόνη πολιτική ε, είναι, μπορούν να είναι αποδέκτες μόνο μιας πολιτικής αλληλεγγύης και ενίσχυσης. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει σε ένα βαθμό. Υπάρχει βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και πιστεύω ότι οτιδήποτε άλλο γίνει θα είναι προ όφελο και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε γιατί σε αυτή την περίοδο κρίσεω βλέπουμε ότι γίνεται μια αναδίπλωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρια υπηρετικά περισσότερο. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρεί την, ε, τα οράματά της στα παγκόσμια και τη φιλοδοξία σε επίπεδο οικουμενικό. Δηλαδή που να καλύπτει και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα, με την, στην έκθεσή μας, επιδιώκουμε να εντοπίσουμε τους, ε, τους φραγμούς εκείνους οι οποίοι δεν επιτρέπουν στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να αντλήσουν κάθε όφελος από την ε, συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν κοιτάξουμε με αυτό το πνεύμα και από πολύ κοντά την κατάσταση, διαπιστώνουμε ότι οι κοινοτικέ πολιτικέ στο σύνολό του έχουν διαγραφεί χωρί να λαμβάνουν υπόψη αυτή την ιδιαιτερότητα και άρα δεν επιτρέπουν την επίτευξη αυτών των στόχων. Επί παραδείγματι, στο περιβάλλον. Μια σειρά κανονισμών μένουν ανεφάρμοστοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές Φερρυπίν και με το πρόγραμμα Horizon 2000, όπου προφανώς εμφανίζεται ανάγκη για ανάπτυξη καλύτερης συνεργατικής σχέσης, αλλά και αντίληψης της ιδιαιτερότητας και των αναγκών των από αποκέντρων περιοχών. Προσπαθούμε λοιπόν να εντοπίσουμε σε κάθε περίπτωση εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα να προταθούν ειδικά ad hoc προγράμματα ώστε να ληφθούν ε, υπόψη οι ανάγκες των πολιτών και των περιοχών, και των, των ε, περιοχών αυτών. Μια νέα προσέγγιση, η οποία πιστεύω στηρίζεται σε μια καλύτερη αξιολόγηση της, ε, α, ε, της ιδιαιτερότητας των από κέντρων περιοχών και που ελπίζω θα τύχει υποστήριξη από όλους τους συναδέλφους. Εάν έχουμε επαρκή χρόνο στη διάθεσή μας, θα ήθελα ιδιαίτερα να εστιαστώ σε μια σειρά από σημεία για να δείξω πόσο μεγάλες μπορούν να είναι μερικές φορές οι αποκλήσεις μεταξύ των στόχων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις οποίες και συμμεριζόμαστε, τους οποίους και συμμεριζόμαστε και τον, τους κανονισμούς και πολιτικών που εν τέλει αναπτύσσονται. Ξέρετε παραδείγματι ότι το ζήτημα της περιφερειακής ενσωμάτωση, καλύτερα ενσωμάτωση των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο περιφερειακό τους περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, είναι γνωστό, άλλωστε αναφέρεται σε όλες τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλην όμως διαπιστώνουμε ότι ε, σε καμία χρονική στιγμή κατά την ε, ανάπτυξη και εκτέλεση των πολιτικών και στο εξωτερικό βέβαια επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξόχως απόκεντρες περιοχές. Το βλέπουμε και στις συμφωνίες εταιρικής, οικονομικής εταιρικής σχέσης ότι είναι πολύ δύσκολο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές να εξασφαλίσουν τη λήψη υπόψη των δικών του συμφερόντων στην ανάπτυξη των πολιτικών. Το ίδιο και στην, ευρωπαϊκή, στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις διαπραγματεύσεις Ε, εξελίξει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Επιτρόπου Ντεγκούχτ και όλων των τρίτων κρατών. Πολύ σπάνια λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των εξόχως απόκεντρων περιοχών ή των προϊόντων τους. Αυτό αποβαίνει των περιοχών ΕΑΠ και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Σε αυτό αποσκοπούν οι προτάσεις μου, ώστε να ληφθούν υπόψη περισσότερο τα ε, συμφέροντα, το, οι ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών. Όσον αφορά τον τομέα της γεωργικής πολιτικής, έχουμε όπως γνωρίζετε ένα ειδικό πρόγραμμα, το λεγόμενο ΠΟΖΕΙ. Ωστόσο διατυπώνουμε προτάσεις επιπλέον για να μπορέσει η γεωρική μας πολιτική να αντλήσει ωφέλη και από άλλα κονδύλια και μέσα, τα οποία ίσως αξιοποιούμε λιγότερο, αλλά που θα μπορούσαν να προσθέσουν ε, περισσότερη αξία ε, στην παραγωγή μας, ε, όπως σε παραδείγματι μια σειρά πιστώσεων και προγράμματα έρευνας. Όσον αφορά λοιπόν την έρευνα και την καινοτομία, μπορούμε νομίζω να εντοπίσουμε ένα σημαντικό πεδίο προς διερεύνηση. Τη, την, ε, τη διαπίστωση αυτή νομίζω ότι συμμερίζονται και άλλοι. Γιατί βλέπουμε ότι τα προγράμματα αυτά, ε, προγράμματα πλαίσιο για την, ανάπτυξη, για την έρευνα και την ανάπτυξη, δεν είναι καθόλου προσαρμοσμένα στην, ε, στις ανάγκες και στις των από αποκέντρων περιοχών. Και εδώ λοιπόν διατυπώνουμε προτάσεις ώστε στον τομέα της έρευνας να υπάρξουν προγράμματα ad hoc, ειδικά προγράμματα με προσαρμοσμένους στόχους που θα αντιστοιχούν στις ετερότες των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Με ένα μόνο παράδειγμα. Όταν, ε, αν ρίξετε μια ματιά στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όλες, πλην ίσως μία, είναι, πλην ίσως η θεστιογενή εδάφη. Ε, κάναμε λοιπόν, ε, έχουμε λοιπόν ε, μια σορευμένη τεχνογνωσία στις περιοχές αυτές. Μια δεξιότητα, θα έλεγα υπεροχή, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος των περιοχών μας στους τομείς της σεισμολογίας, ηφαιστειολογίας, γενικά φυσικών καταστροφών, αλλά και προς όφελος ταυτόχρονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πρόκειται για ζητήματα που ασφαλώς αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι καταλάβατε τι επιδιώκω με την έκθεση. Και να συνεχίσω αυτήν την πολιτική της αλληλεγγύης και της κάλυψης του χαμένου εδάφους, αλλά και να στηρίξω τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στην ε, αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες και να δείξω ότι οι επενδύσεις σε αυτές τις εξόχως περιοχές είναι επενδύσεις ωφέλιμες και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. του λεχθέντος και σταματώ εδώ προς το παρόν. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν αποκλειστικά και μόνο εάν χορηγήσουμε τη θέση που του αρμόζει στο άρθρο 349 εάν αναγνωρίσουμε τη σημασία και τη θέση του άρθρου 349 για το σύνολο των πολιτικών που αναπτύσσει και υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια νοοτροπία σχετική με το άρθρο 349 σε επίπεδο Γενικής Διευθύνσεως των Περιφερειακών Υποθέσεων. Ασφαλώς και κάποια νοοτροπία σε επίπεδο της Γενικής Διευθύνσεως γεωργίας που το χρησιμοποιούν ήδη, αλλά δεν υπάρχει επαρκής νοοτροπία και αναγνώριση της σημασίας του 349. Θα λέγω ότι είναι ελλειπής η αξιοποίηση του άρθρου αυτού στις λοιπές γενικές διευθύνσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί μπορεί το 349 να ενταχθεί στην, ε, στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι για να αποτελούμε μια διαρκή παρέκκληση στους στόχους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για να εξασφαλίσουμε χάρη στο άρθρο αυτό στις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές μας να επιτύχουν τους στόχους που ορίζει σύν το χρόνο βεβαίως τους στόχους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω οι προτάσεις σας να εμπλουτίνουν την έκθεση με τις τροπολογίες σας. και περιμένω πολλά από τη συζήτηση που θα γίνει σήμερα για να ενισχύσουμε τη διατύπωση των πρώτων αυτών προτάσεων που συζητούμε για πρώτη φορά σήμερα το πρωί. Εμεί ευχαριστούμε. Και τώρα, οι σκιώδες Πρώτα πρώτα του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον εισηγητή Γιούνου Μαζί για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ε, πιστεύω ότι είναι πολύ καλό παράδειγμα αγαστής συνεργασίας ε, βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προέρχονται από εξόχως από κέντρες περιοχές. Ε, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν αυτής της συνεργασίας κατά την τρέχουσα θητεία. Ε, επίσης ε, καταδεικνύεται η ιδιαίτερη σημασία που προσδίδει ιδιαίτερα η Επιτροπή μας και γενικότερα το Κοινοβούλιο σε αυτές τις περιοχές κυρίως ως προς ε, αυτά που θα κληροδοτήσουμε στους βουλευτές της επόμενης κοινοβουλευτικής θητείας για το κοινοτικό κεκτημένο, αν θέλετε, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Βλέπουμε τη δυνατότητα δημιουργία ε, συνεργειών ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία και των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, μέσα αυτή την εκθεσία ο συνάδελφος ο Μαρζή κάνει διάφορες προτάσεις, ιδιαίτερα εύστοχες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Από πλευρά μου το μόνο που θα αποπειραθώ να κάνω είναι να συμβάλλω κι εγώ στη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ε, πιο συγκεκριμένα, η ομάδα των βουλευτών που επεξεργάστηκαν αυτήν την έκθεση όπως εξήγησαν και σε διάφορες άλλες συναφείς εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε διάφορα άλλα έγγραφα των σκιωδών εισηγητών που απίφθηναν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι και εγώ ε, θα καταθέσω διάφορες συμπληρωματικές τροπολογίες που στόχο έχουν ε, πολύ συγκεκριμένα το εξή. Πρώτα απ' όλα να επιμείνουμε στη σημασία των ε, μακροπεριφερειακών στρατηγικών για την εξαιρετικά εργαλεία δημιουργίας ε, νέων συμπράξεων και χαρακτηριστικά παραδείγματα προσέγγισης όπου εμπλέκονται πολλά ταμεία. Ε, επίσης, ε, ε, προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις δημόσιες υπηρεσίες κοινή ωφέλειας, κυρίως για την ενημέρωση, τις τηλεπικοινωνίες, για τις μεταφορές και την ενέργεια. Ιδιαιτέρως τονίζουμε την καταλητική σημασία που έχουν οι επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών για τις εξόχως από κέντρες περιοχές. Η Επιτροπή ε, μας ούτως ή άλλως έχει προτείνει πολλά σε προγράμματα όπως το ΠΟΖΕΙ ε, για να ε, προωθηθούν οι μεταφορές. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο Εράσμους και στο Εράσμους Μούντους και τις σχέσεις μπορούν να υπάρξουν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πέρα από την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση ε, στη χρηματοδότηση για να πραγματοποιηθούν άλλες επενδύσεις. Θα στηρίξουμε και τις πρωτοβουλίες αυτών των περιοχών για την απασχόληση των νέων και τις επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για τους νέους. Όπως μας είπε ο εισηγητής, θα πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα ΠΟΖΕΙ ε, και ε, το ΠΟΖΕΙ για τη γεωργία και την αλληλεία ε, είναι τομείς που είναι καθοριστική σημασίας για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών για το ΠΟΖΕΙ αλία ο εισηγητής δεν αναφέρθηκε ίσως επαρκώς στον γενικό κανονισμό για την αλλία για τους ελέγχους Ε, όπως τόνισαν οι βουλευτές που προέρχονται από τέτοιες ε, περιοχές, ε, πρόκειται για ένα αναφέρετο δικαίωμα των περιοχών να συμμετέχουν ισότιμα στις βασικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Να τον συγχαρώ και πάλι για την εξαιρετική ποιότητα της έκθεσής του. Θεωρώ ότι θα επηρεάσει δε σε σημαντικό βαθμό τις μελλοντικές πολιτικές που θα επηρεάσουν στις εξόγους από περιοχές. Θα θα ήθελα κλείνοντας να δηλώσω την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε περαιτέρω με τους συναδέλφους και κλείνοντας να διαβάσω όπως ε, ένα κομμάτι της έκθεσης ε, βλέπουμε ότι οποιαδήποτε επιτυχία σημειώνεται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι θρίαμβος για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτή η φράση πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους, ε, διότι θα πρέπει να κοιτάζουμε ψηλά προς τον ουρανό αν θέλουμε να εισακουστούν οι προσευχές μας ε, και όχι να σκύβουμε το κεφάλι μόνο, έτσι θα εξασφαλίσουμε την επιτυχία. Ευχαριστούμε ο Σεπάολο Αλβεσέ ε, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι ήδη αναφέρθηκαν όπως και ο εισηγητής στις βασικότερες συνιστώσεις και βασικότερες προκλήσεις που υπάρχουν για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές κυρίως για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στον Ατλαντικό ή ε, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας και τα υπερπόντια εδάφη της που ε, εκτείνονται μέχρι και την Βόρεια Αμερική. Αφρική, τον ε, Ινδικό ωκεανό και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ικανοποιητική συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής. Ο στόχος είναι η βελτιστοποίηση κατάστασης αυτών των περιοχών, δημιουργώντας συνέργειες ανάμεσα ε, στα διαρθρωτικά ταμεία και τις, ε, τα υπόλοιπα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζεται ότι πρόκειται για θρίαμβο τη Ευρωπαϊκής Ένωση η πρόοδος των από απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης που είναι και σημαντικότερη πρόκληση για όλους και βλέπουμε ότι ε, στον τομέα των επιστημονικών, των κλιματικών αλλαγών, ε, στον τομέα των ε, πλούτοπαραγωγικών ορεικτών των ε, ε, πλουτοπαραγωγικών πόρων πιο συγκεκριμένα κτλ. κτλ ε, μπορούν να, σημειωθούν, να σημειωθεί μεγάλη πρόοδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των εξόχως από κεντρών περιοχών. Το ίδιο ισχύει για όλες τις περιοχές δε, όπου και αν βρίσκονται αυτές. Και πιστεύω ότι ε, όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να επωφεληθούν από τέτοιες ε, δράσεις ε, Πιστεύω ότι κάποιε πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν καθοριστική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσουν. Ναι, κυρίω να τονίσουμε τη σημασία συγκεκριμένων οργάνων και εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν όλου ιδιαίτερω σε αυτέ τι περιοχέ. Ε, Παραδείγματο χάρη Ευρώπη 2020, Ενεργεία 2020, Life, Erasmus, προγράμματα στον τομέα τη ενέργεια των τηλεπικοινωνιών μεταξύ άλλων. Αυτές οι πολιτικές και αυτά τα εργαλεία στην εφαρμογή τους ε, θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών ε, ούτως ώστε να εκπληρώσουν στο έπακρον τον στόχο που έχει προκαθοριστεί και να εξασφαλίσουν ε, ισότιμα επίπεδα ανάπτυξης για αυτές τις περιοχές όπως και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Βλέπει ο εισηγητής στην έκθεσή του περαιτέρω δυνατότητες βελτίωση της χρήσης αυτών των εργαλείων ε, και νέων συνεργειών ανάμεσα στι επιμέρου πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση και των διαρθρωτικών ταμείων υπάρχει, ε, υπάρχουν επίση άλλε συνιστώσει των ε, εφιστάμενων πολιτικών που μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω και κυρίω μέσα από μια καλύτερη συνεργασία μπορούμε να αναπτύξουμε τι ιδιαίτερε δυνατότητε και ιδιαίτερο δυναμικό που έχουν αυτέ οι περιοχέ και να καταπολεμήσουμε τι αδυναμίε του. Και ξαναλέω ότι οποιαδήποτε πρόοδο σημειωθεί σε αυτέ τι περιοχέ περιοχές θα είναι υποφελής για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν μέχρι το τέλος της ε, πρώτης εβδομάδας του Ιανουαρίου να παραταθεί η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών ε, και όχι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, τόσο ώστε με το που ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας τον Ιανουάριο να έχουμε αρκετό χρόνο να επεξεργαστούμε αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you. For Greens we have Jean-Jacques I think he's not here, right? Mm-hmm. Επίση και ο διοικητή είναι ο Ζων Ζόγκμπιση, αλλά δεν υπάρχει το σε κάποιο να τον καταστήσει. Όχι, επομένω ε, έχουμε τώρα την συζήτηση. Πρώτο είναι ο κύριο Νίλσον. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά αφού μου δίνετε τη δυνατότητα. Αυτή η έκθεση είναι πάρα πολύ. Καλή ποιότητα και ιδιαίτερα επίκαιρη, διότι ε, πραγματεύεται διάφορα ζητήματα, τα οποία πρέπει να μα απασχολούν σε όλες ε, τις ε, περιοχές. Με ποιο τρόπο μπορούμε να συντονίσουμε τι δράσει των διαρθρωτικών ταμείων με άλλε πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βόρεια Σουηδία, από όπου προέρχομαι εγώ, τίθεται αυτό το ζήτημα. Ποια είναι η στρατηγική των περιοχών, ώστε να επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό όλων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Και το αφήνουν όλοι στα χέρια των περιοχών περιφερειών. Πρέπει να επιλύσουν αυτό το δύσκολο πρόβλημα. Η πρόεδρος, η κυρία Χίμπνερ, ε, θα, ε, σωστά μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε η πολιτική συνοχή σε πώς θα μετατραπεί σε ένα εργαλείο τόσο ώστε να εφαρμοστούν καλύτερα οι υπόλοιπες τομιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στον Βορρά και στον Νότο και το, η σημαντικότερη πρόκληση είναι ο καλύτερος συντονισμός. Και αυτό είναι το βασικό ζητούμενο για μένα αλλά και για τον εισηγητή. Εγώ θεωρώ ότι η βασική μας μέρημνα θα πρέπει να είναι οι εθνικές αρχές, δηλαδή οι περιφέρειες προσπαθούν να βρουν τις διάκριτες γραμμές ανάμεσα στα διάφορα ε, επιμέρους προγράμματα ε, και να υπερβούν αυτά τα σύνορα. Ε, και αντίθετα οι εθνικές αρχές χτίζουν νέα τείχη που χωρίζουν τις περιφέρειες και χωρίζουν τα επιμέρους προγράμματα και καθιστούν αδύνατο τον συντονισμό. Θα έπρεπε Πρέπει λοιπόν μέσα στην έκθεση να τονίσουμε ότι θα πρέπει να ε, απευθύνουμε επικριτικά σχόλια κατά των εθνικών αρχών. Δεν πρέπει να περνάμε το μήνυμα ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τη δράση των εθνικών αρχών. Ε, ευχαριστώ, λίγο, Πρόεδρος. Δεν είμαι σκιώδης εισηγήτρια. και μόλις τώρα έριξα μία ματιά στην έκθεση αλλά επισήμανα κάποια ενδιαφέροντα σημεία ιδίως εκεί που μιλάει για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί και εγώ είχα συμμετάσχει στην ισομερή συνέλευση με τις χώρες ε, ΑΚΕ και ε, είναι θέμα το οποίο ανακύπτει παγίως και συνεχώς σε σχέση με τις χώρες εκείνες που είναι και ε, εξόχως κεντρες ε, περιοχές και πρόκειται για τους πόρους επομένως που αποτελούν κάποιο τρόπο το μήλο της έρηδος. ή πολλέ φορέ τέλο πάντων, ενώ τα πάμε καλά σε, σε άλλου τομεί, εκεί υπάρχουν προβλήματα. το Σουρινάμ, ε, ήταν το θέμα εκεί των ε, συνόρων. Ε, είχαμε διάφορους οι οποίοι μπαίναν από το Σουρινάμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν εύκολο και είχε θεωρηθεί ότι η αστυνόμευση, η φύλαξη εκείνων των συνόρων ε, ήταν δύσκολη με τη θεωρία διαβατηρίων, τα διαβατήρια κλπ. υπήρχε θέμα. Οπότε θα πρέπει σε σχέση με αυτά που σα επισήμανα θα κατεβάσω κάποιε τροπολογίε. Αλλά καταρχήν συμφωνώ και θα τα ξανασυζητήσουμε ίσω και σήμερα ότι θα πρέπει κάπω να τονιστεί περισσότερο το ότι δεν έχουμε αρκετή βοήθεια από εμπειρογνώμονε στην ε, Επιτροπή μας. Δεν, δεν, δεν έχουμε τις ειδικές γνώσεις εμείς. Ε, επίσης όσον αφορά κινήσεις πληθυσμών, γεωργία, εμπόριο ότι πιο όλα αυτά εδώ ε, ανακύπτουν. Άρα θα έπρεπε να το ξαναδούμε το τι θα κάνουμε με τις εξόχους αποκέντρες περιφέρειες εδώ στην ε, Επιτροπή μας. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Εάν όχι, ο εισηγητής να απαντήσεις σε όσα άκουσε. Σας ευχαριστώ. Ναι, να σας πω, ε, ξεκινώντας από την τελευταία, συναντού που το λόγο. Τα προβλήματα των από κεντρών περιφερειών και περιοχών είναι προβλήματα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι θέματα ε, όχι μόνο περιφερειακής πολιτικής αλλά όλων των πολιτικών γιατί βλέπετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν όσον αφορά την στρατηγική για τις εξώσεις από τις περιοχές ήταν ζητήματα που έχουν απασχολήσει όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου, όλες τις ε, γενικές διευθύνσεις της ε, Κομισιόν. Άρα θα πρέπει να κινητοποιηθούμε περισσότερο όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ όλους τους ε, αγορητές για τα όσα είπαν και θα δούμε ένα-ένα τα όσα προτάθηκαν και να απαντήσουμε σε μία-μία τις ερωτήσεις. Αναφέρθηκε το πρόβλημα του ότι δεν έχουμε πια το ποσεή για την αλία και το ότι υπάρχουν τώρα φόφοι φόβοι σε σχέση με την τύχη που θα έχει το ΠΟΣΕΗ για την γεωργία. Και ε, το είπα στο τέλος της ε, εισήγησής μου ότι δεν ξεχνούμε πως το ΠΟΣΕΗ είναι τεράστια σημασία. Και βεβαίω το άρθρο 349 της συνθήκης για την κοινή αλληλευτική πολιτική ε, είναι συγκεκριμένο μέσο πολιτικής αυτό, συγκεκριμένο εργαλείο το, πόση, το πρόγραμμα πώς για την αλληλεία. Δεν συζητάμε τώρα για περιεχόμενο κάποιων μέτρων, μιλούμε τώρα για το τι πολιτικό μήνυμα θα, θα στείλουμε Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν ανησυχίες, δηλαδή θα πρέπει να συμπεριληφθούν και να καλυφθούν περισσότερο οι από τις περιοχές της κοινωνικής πολιτικής. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο χαλαρότητας εφαρμογής του άρθρου αυτού. Βεβαίω και κατά τα λοιπά θα πρέπει να κάνουμε και άλλες προτάσεις όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Και εδώ είναι θέμα σοβαρό, επί το οποίο θα υπάρξουν και άλλες τροπολογίες. Ο Λουίς Άλβες μας μίλησε για την ε, παγκόσμια διάσταση που μας φέρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ε, ε, η κάθε από κεντρη περιφέρεια και περιοχή. Ναι, το χρειάζεται συντονισμό της στρατηγικής μας. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι πολύ χρήσιμες οι σχετικές ε, τροπολογίες. Εμεί όλοι που ερχόμαστε από αυτέ τι περιοχέ θα πρέπει να συναντηθούμε και από κοινού να κατεβάσουμε κάποιε τροπολογίε ακριβώ όπω ετώνησα ε, ε, στου ε, συναδέλφου τη Επιτροπή μα ότι είμαστε μια ομάδα που προέρχεται από τι εξόχου κεντρικέ περιοχέ και πέραν τη κομματική προέλευση συνεργαζόμαστε συνεχώ, ούτως ώστε να μπορούμε να εισφέρουμε με κάποιες προτάσεις ε, για τις ε, περιφερειές μας. Και επαγρυπνούμε για τα συμφέροντα αυτών των περιφερειών εδώ από το μετερίζου του Κοινοβουλίου. Επίσης, κάτι άλλο που αναφέρθηκε και είναι σημαντικό, οι σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Κοιτάξτε τι προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε. τα υπερπόντια εδάφη διαμερίσματα, οι χώρες ΑΚΕ. Θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλη συνάφεια μεταξύ των προβλημάτων των, που έχουν οι μεν και οι δε. Υπάρχει αντιστοιχία, υπάρχει παραλληλισμός γιατί οι περισσότερες από τις χώρες ΑΚΕ είναι μικρά νησιωτικά κράτη, αναπτυσσόμενα και έχουν επομένως τα ίδια προβλήματα που έχουν και οι από τις περιφέρειες. Οπότε έχουμε θέματα, προβλήματα ε, ενεργειακής πολιτικής, προβλήματα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, προβλήματα δημογραφικά, προβλήματα που προκύπτουν από την νησιωτική φύση, από το, τροπικό τους κλίμα, κοινά επόμενα τα προβλήματα, κοινά τα διακυβεύματα, οι προκλήσεις, οπότε τι πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει στις εξόχους από τις περιφέρειες είναι επίσης βάση και εμπειρία για να παρέμβει κανείς, να βοηθήσει κανείς αυτά τα, άλλα κράτη τα οποία είναι τόσο συναφή με τις εξόχους από τις περιφέρειες. Ε, Επίσης αυτό ισχύει και για τα περιποντία διαμερίσματα. Και εκεί υπάρχει συνάφεια και εκεί υπάρχουν ομοιότητες πέραν των νομικών διαφορών. Βιοπικιλότητα, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πολιτιστική πολυμορφία, βέβαια όλα αυτά ισχύουν, αλλά κατά τα άλλα Υπάρχουν ε, πάρα πολλά κοινά σημεία όσον αφορά τα αντιμετωπιζόμενα προβλήματα. Ε, τα λέμε αυτά στην έκθεση, ότι θα πρέπει όσο είναι δυνατόν αυτό να αναδείξουμε εδώ με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να προκύψουν κάποια προγράμματα τα οποία να καλύπτουν τις εξώχους απόκεντρες περιφέρειες αλλά και τα και διαμερίσματα. Σημαντικό, γιατί το Συμβούλιο. Δεν εκπροσωπούνται οι εξόχους από τις περιφέρειες. Εκπροσωπούνται μόνο από τρεις χώρες, τρεις χώρες μέλη. Γαλλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Με τα δε διαμερίσματα κάπως αυξάνεται η επιρροή που μπορούμε να έχουμε στο, στο Συμβούλιο. Και έτσι έχουμε κάπως περισσότερο ειδικό βάρος στο Συμβούλιο. Πάει το ζήτημα της μετανάστευσης, τα προβλήματα τα συγκεκριμένα της ε, Γουιάνας και της Μαγιώτ. Υπάρχουν και κάποιες αντιφάσεις οι οποίες προκύπτουν όσον αφορά τη φτώχεια. Οπότε είναι σημαντικό θέμα η ανάπτυξη γιατί υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες δυσκολίες που είναι δύσκολο να τις ε, διαχειριστεί κανείς. Και η πολιτική μετανάστευση που ασκείται στην υπηρετική Ευρώπη δεν αντιστοιχεί και δεν ισχύει ε, αναγκαστικά στις νησιωτικές εκείνες ε, περιοχές. Αυτά οπότε με τις προτάσεις που έχουν ε, διατυπωθεί πιστεύω ότι θα μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας η οποία να είναι πραγματικά φιλόδοξη, να εμπίπτει στους στόχους μας και που να καταλήξει τελικά σε κάποια καινούργια προγράμματα τα οποία θα αρχίσει να τρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία θα είναι προσυρμοσμένα και θα αντιστοιχούν με τις ανάγκες που έχουν οι εξόχους απόκεντρες περιφερειές μας. Πρόεδρος Γιούνος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τροπολόγια ε, θα έχουμε ως ε, προθεσμία ε, την 7η Ιανουαρίου. Μέχρι την 7η Ιανουαρίου το μεσημέρι μπορεί να υποβάλλετε τις τροπολογίες. Οπότε τώρα τελειώνει αυτό το σημείο τη διατάξεω και πάμε εις τις ψηφοφορίες. Αλλά περιμένουμε ακόμα ένα λεφτάκι να έρθει ο κόσμος. Αλλά στο μεταξύ μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν δουλεύουν οι κάρτες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν θέλετε δοκιμάστε, βάλτε τις κάρτες να κάνουμε τη δοκιμή. Ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Try to vote now so we can see what... Συνάδελφοι, προσπαθούμε να ψηφίσουμε δοκιμαστικά το να δούμε αν δουλεύουν οι κάρτες. Ah, it, was not here in a second, a second ago. Okay, that's perfect. It should work now, yeah. should work, yeah, works, I think five colleagues didn't check. Yeah, you're moving. Okay, so I, think we can close the... Α, ωραία, εντάξει. Άρα να θεωρούμε ότι έληξε η ψηφοφορία. Και πάμε τώρα στην πρώτη ψηφοφορία της μέσης διάταξης. A situation where we need your, the information from you, you tell us how you voted, right? Uh, are you sure? Α, ξέχασες την κάρτα. Καλά, πες μας τότε τι ψηφίζεις, αν χρειάζεται. Ξεκινούμε με την έκθεση Σρέντερ. Συμβαστική Β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 είναι γλωσσικό το θέμα, θα ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 γλωσσικού χαρακτήρα εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 εις δύο τμήματα το πρώτο υπέρ Έλέγχο του αποτελέσματο στο 24 πρώτο τμήμα πέρας και εγκρίνεται τώρα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ και τώρα κάνουμε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται Συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 ε, και 38 είναι ταυτόσιμες. P είναι υπέρ. Πώς? Α, παρέλειψα την 29 λέει η κυρία Χούμνερ Την 28. Παρέλειψα την 20. Α, συγγνώμη, συμπαθάτε με, λέει ο πρόεδρο. Ξαναγυρίζουμε. Πίσω πάμε στο 28. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Η 30 καταπίπτει. Συμβαστική J ψηφίστηκε. 37 και 38 υπέρ. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική κάπα καταπίπτει. Ελ. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Ναι. Ψηφίζουμε το L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, συγγνώμη, είναι ακόμα πρωί και κοιμάμαι γιατί εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Η ΕΛ επομένω έχει δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα του ΕΛ. Υπέρ. Έλεγχο για το πρώτο τμήμα του ΕΛ. Εγκρίνεται. Και τώρα θα πάμε στην ε, τροπολογία 45, αν δεν κάνω λάθος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N εις δύο τμήματα. Το πρώτο του N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα έλεγχος για το δεύτερο τμήμα του N. Πέρας και εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Ψηφίζουμε το 53. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53. Έλεγχος, όπως ζητήθηκε από τους συναδέλφους. Έλεγχος για το 53. Πέρας. Εγκρίνεται. 25, 54 καταπίπτει και πάμε στη συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Π. Συμβαστική π. Πρώτο τμήμα μόνο το πρώτο Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 60. Τροπολογία 60. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κωνσταντς, ψηφίσεις κατά της τροπολογίας σου. Α, πρέπει να κάνω έλεγχο. Έλεγχος για το 66. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις βιβλικές παραγράφους. Ε, τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική 2. Υπέρ κατά ε, ε, συμβαστική α για τις αιτιολογικές. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική π. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα. Ήτρε. Η παριθμόν 1 καταπίπτει. 2 ε, ε, πάμε στο 3. Ψηφίζουμε το 3 της Ήτρε. Υπέρ. 3, 3. Τροπολογία. Α, καταπίπτει και αυτή. Λάθος. Μου είπαν ότι πάμε στο 4. Εδώ η, η επαΐουσα λέει ότι πρέπει να, ψηφίσουμε το 4. Και το κάπα δεν ψηφίστηκε, δεν εγκρίθηκε, υπέρ καταποχής δεν εγκρίνεται. 5 ήτρε υπέρ, κατά, έλεγχος για το 5. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της ήτρε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 κατά διέρεση εδώ η χωριστή ψηφορία το πρώτο καταπίπτει το δεύτερο το δεύτερο του 7 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα εγκρίνεται και οι 8 και 9 καταπίπτουν και πάμε στο 10 υπέρ υπέρ έλεγχος για το 10 ψηφίζουμε πέρας εγκρίνεται το 11 καταπίπτει όχι πρέπει να το ψηφίσουμε το 11 γιατί απερίφθη το K. έλεγχος ηλεκτρονικός για το 11 ψηφίζουμε πέρας Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα. Ποια θα ψηφίσουμε. 18. Ψηφίζουμε την 18. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ έλεγχος για το 20. Ψηφίζουμε πέρας. Εγκρίνεται το 20. Το 21 καταπίπτει. Το 22 επίσης. 23 υπέρ. Κατά. Ο έλεγχος για το 23. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέραση εφορίας 32 υπέρ εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Και πάμε τώρα στο σημείο 6. Είναι η έκθεση. Η έκθεση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ... Ας επαληθεύσουμε την τροπολογία 7 παρακαλώ. Πέρας στην 8 προφορική τροπολογία είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας όχι. Δύο τμήματα. Όπως τροποποιήθηκε το ψηφίσαμε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 2 της Επιτροπής των Προϋπολογισμών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ελέγχουμε τη 2 των προϋπολογισμών πολύ καλά πέρασε ομόφωνα. Ποιος τι θέλει να ελέγξουμε. Ελίζα Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 6 των προπολογισμών υπέρ. 6. 13, 14 και μετά η 6 λαμπέ. Τον έχω τον καταλογό σα είναι εκεί πέρα. Έξι των προπολογισμών και το ΕΛΚ είναι υπέρ, το έχω. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 προφορική. Δεν υπάρχει κανεί. Ε, δεν αντάσσεται κάτι, κανείς την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 16 επίση με προφορική, υπάρχει καμιά αντίρρηση, όχι, την ψηφίζουμε όπω τροποποιήθηκε, υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 19 μα είσαι πολύ γρήγορη σήμερα 19 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ επαληθεύουμε την 22 άρχεται ψηφοφορία Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ 17 κατά, 23 με προφορική, υπάρχουν αντιρρήσει όχι, την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 26-27 μαζί υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 με προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις όχι, ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Ας επαληθεύσουμε την 35, 35 επαλήθευση. Πέρας. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απερίφθη. 22 κατά 17 υπέρ. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 πεσύρθη, 45 προφορική, υπάρχει αντίρρηση, όχι, την ψηφίζουμε με προφορική τροπολογία, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 48, πάλι με προφορική τροπολογία, υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι, την ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 και τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις όχι όπως τοποποιήθηκε λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 55 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 56 τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 59 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 68 προφορική τροπολογία, υπάρχει αντίρρηση όχι, όπως τροποποιήθηκε λοιπόν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική έτσι 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 69 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 78 με προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι υπέρ λοιπόν, όπως προπήθηκε κατά αποχές εγκρίνεται, 79 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 με προφορική παλιτροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις όχι, όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 πάλι με προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις όχι όπως τροποποιήθηκε λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και στις αιτιολογικές ε, προτάσεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο υπέρ κατά αποχές απερίφη τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ υπάρχει ψηφοφορία Πέρασε. 35 πέρα μία ψήφο κατά τρει αποχές, εγκρίνεται συγχαρητήρια. Και πάμε στην ε, γνωμοδότηση Γιώαχιμ Τσέλερ. Υπαριθμόν ανατροπολογία υπέρ, κατά απόχε. εγκρίνεται. Δύο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ, κα, υπέρ. Τροπολογία 3. Κατά αποχές απερίφθη 1 συμβαστική 1 υπέρ Α, με συγχωρείτε, προφορική τροπολογία στη συμβαστική 1. Ε, υπάρχουν αντιρρήσει η Κωνσταντσα. Μάλιστα. Άρα την ψηφίσουμε χωρί τη, συμβαστική, χωρίς τη ε, πρόσθετη προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Στη συμβαστική 2 επίση με προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσει. Πάλι Κωνσταντσα. Κρέλ, υπέρ, χωρίς τροπολογία λοιπόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην υπαριθμόν 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 11 με προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Ουδής, άρα την ψηφίζουμε με τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Επαληθεύουμε τη 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Αρ. Μιγγέλ. Ναι, ξέρω, σήμερα ο Μιγγέλ κοιμάται. Έχουμε λοιπόν στη 16 σε τμήματα παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο δεύτερο τμήμα υπέρ επαληθεύουμε ηλεκτρονικά Δεύτερο τμήμα. Πέρες ψηφοφορία. απερίφθη 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειονοψηφία και περνώ στην κυρία Λούκα Τσαιέσκα. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση. Αρχίζουμε. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ επαληθεύουμε την 8 αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε 25 υπέρ, 13 κατά υπέρ, 9 ε, παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, αιτιολογικές σκέψεις, ε, τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κα... Με συγχωρείτε. Α, καταπίπτει, συγγνώμη. Δεν χρειάζεται να εκφραστείτε κατά. Συμβαστική 6 λοιπόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κα, συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 παρακαλώ υπέρ. Επαληθεύουμε την τροπολογία 4. Πέρασε προφορίες Εγκρίνεται 21 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία. Αρχίζει παρακαλώ. Πέρασε. Με μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τις προφορίες μας. Και παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι να μείνετε στην αίθουσα, διότι πρόκειται να, γίνει, να ληφθεί μια πολύ σημαντική απόφαση. Έχουμε να εγκρίνουμε μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη που συζητήθηκε, αναφέρθηκε στην αρχή της συνεδριάσεως. Μετά τις προφορίες λοιπόν προσθέτουμε ένα νέο σημείο σχετικό με μια απόφαση του Συμβουλίου για πρόταση της, Ευρωπαϊ... πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύτερα για απόφαση του Συμβουλίου, γιατί σε αυτό το στάδιο βρίσκεται η νομική διαδικασία, ε, που επιτρέπει στη Γαλλία να επιβάλλει μειωμένο ε, συντελεστή έμεσου φόρου για το ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάννα και την Ρεουνιόν. Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά το έτος αυτό και μετά και όπως ε, στο παρελθόν για τις Κανάριες νήσους πριν από μερικές μήνες συγκεκριμένα όταν δεχθήκαμε τη διαδικασία της ε, διαβούλευσης, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είπαμε ότι μπορούν να, γίνουν παρεκκλήσεις για πολλά προϊόντα για, των Καναρίων από αυτή την ε, αυτοσυντολιστή εμέσου φόρου με βάση τη διαδικασία του άρθρου 46, απλουστευμένη διαδικασία και μπορούμε έτσι να κάνουμε την ίδια διαδικασία και εδώ και να λάβουμε σήμερα την απόφαση. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τεχνικού χαρακτήρα απόφαση, όπως και με τα Κανάρια. Επεκτείνουμε δηλαδή υφιστάμενους κανόνες. Επεκτείνουμε το πεδίο υφισταμένων κανόνων. Μπορώ να σας δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες αν θέλετε. Ε, πρόκειται για μια απόφαση η οποία θα επιτρέψει τη Γαλλία στο παραδοσιακό αυτό ρούμι που παράγεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της και που πωλείται στην υπηρετική Γαλλία, στην υπηρετική επικράτεια της Γαλλίας, να επιβάλλει ένα μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης και να απελευθερώσει αυτά τα προϊόντα, να απαλλάξει τα προϊόντα αυτά από ένα ειδικό φόρο που σχετίζεται με ένα ειδικό ταμείο, που πηγαίνει σε ένα ειδικό ταμείο για συγκεκριμένε ασθένειε, χρηματοδοτεί την αντιμετώπιση κάποιων ασθενειών. Έτσι λοιπόν, ετήσια ποσόστοση για το ε, πολλούμενο στην ε, πυρωτική Γαλλία Ρούμι αφορά, επίσης αφορά μια και προβλέπει μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Το 2017 δηλαδή η Γαλλία θα κληθεί να ε, καταρτήσει μια μεσοπρόθεσμη έκθεση με την οποία θα δείχνει αν υπάρχει λόγος και ανάγκη να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς της παρέκκλησης ή αν υπάρχει πλέον, έχει πλέον εκλείψει ο λόγος για την έκτακτη υποστήριξη για το ρούμι από ζαχαροκάλεμο που παράγεται στις από απόκεντρες περιφέρειες της Γαλλίας η κατάσταση λοιπόν είναι αυτή η ισχύουσα νομοθεσία εκπνέει τώρα το Δεκέμβριο Δυστυχώς και λόγω καθυστερήσεων στις εργασίες του Συμβουλίου η απόφαση αυτή φτάνει με μεγάλη καθυστέρηση στο Κοινοβούλιο και δεν μπορέσαμε να την δούμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Άρα ούτως ή άλλως μόνο τον Ιανουάριο μπορεί να τον εγκρίνει η Ολομέλεια του σώματος, αλλά αυτό δεν οφείλεται σε κάποια ε, του Κοινοβουλίου. Οφείλεται στην καθυστερημένη υποβολή της προτάσεως από το Συμβούλιο. Το μόνο μπορώ να πω σε αυτό το στάδιο είναι ότι μπορούμε μέσω του άρθρου 46 να αποφύγουμε την συνήθη διαδικασία των τροπολογιών και των συζητήσεων της εκθέσεως και όπως έγινε και με τα Κανάρια να δώσουμε την άδεια στην Πρόεδρο της Επιτροπής, εφόσον εσείς βέβαια το εγκρίνετε σήμερα, για την, προ... για την ε, περαιτέρω πρόοδο στη διαδικασία αυτή τη διαβούλευση. Να σα πω επίση ότι πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία το Συμβούλιο μπορεί να μα αγνοήσει. Δηλαδή η διαδικασία των διαβουλεύσεων ή θα ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο ή μπορεί και να μην ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο, δεν είναι υποχρεωτικό. Πάντως πρέπει εμείς να την ολοκληρώσουμε. Αυτά έχω να πω προ το παρόν. Μπορούμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε το 46 με την απλουστευμένη διαδικασία ή αλλιώς θα ακολουθήσουμε την πλήρη νομοθετική διαδικασία. Πράγμα βέβαια το, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε έτοιμοι για τη σύνοδο του Ιανουαρίου. Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς τώρα. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι η Κατρίν Μπέτερ έχει ήδη επισημάνει το θέμα αυτό και θέλω να της δώσω το λόγο γιατί θέλει να εκφράσει τις επιφυλάξεις και τους δισταγμούς της για το θέμα αυτό. Κατρίν. Ήδη συζητήσαμε το τον εξόχως από ματισμένο περιοχών και όπως είπες δεν θα μπορούσαμε να πούμε να κάνουμε και πολλά γνωμοδοτούμε και μπορεί και να μην ληφθεί υπόψη αυτό που θα πούμε. Πάντως, νομίζω ότι το θέμα είναι ότι με αυτές τις ρυθμίσεις με το Ρωμί έχουμε στρέβλωση της αγοράς στη Γαλλία. Οπότε είναι θέμα ενιαίας αγοράς και όχι τόσο θέμα εξόχως από περιχών. μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν είχαμε την ευκαιρία να προβούμε σε αυτή την αναθεώρηση των όρων και προϋποθέσεων, οπότε ενδεχομένως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κατά πόσον είναι δική μας αρμοδιότητα και να δούμε πώς το μέλλον θα διαχειριστούμε αυτές τις εκθέσεις. Εγώ δεν είμαι κατά το, το, το, να φροντίσουμε τις ειδικές ανάγκες των περιφερειών αυτών, όπως είπαμε, αλλά το 60% της ζάχαρης στη Μαρτινίκα γίνεται ε, ρούμε στη Μαρτινίκ και 40% στην ε, Γουαδελόπη Είναι ε, πολύ ρούμι αυτό και γι' αυτό και φέρνει στρέβλο στην αγορά. Οπότε μπορεί να ξανακαταλήξουμε στο, στο, στο, στο, θέμα εκείνο, στην πολεμική, όπως έγινε με την μπανάνα. Δεν θέλουμε να επαναληφθεί αυτό, αλλά όμως έχουμε πάρα πολλούς παραγωγούς ε, ρουμιού στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πρόβλημα. Δεν έχει νόημα να απορρίψουμε την έκθεση, γιατί έτσι καλώς πρέπει να έχει περιοθεί, αλλά να δούμε στην επόμενη θητεία τι θα κάνουμε με τέτοιες εκθέσεις. είναι σχεδόν ύβρις, είναι σχεδόν προσβλητικό αυτό, γιατί μας παρακάμπτουν ουσιαστικά, Πρόεδρος. Ναι, να δούμε με ποια διαδικασία θα προχωρήσουμε, όπως συζητήσαμε, τέλος με την Κωνσταντσα και για τον Γιάνν Άλμπρεκτ, Κωνσταντσα και για τον Γιώργο μαζί. Ευχαριστώ πολύ, Ντανούτα. Δεν είναι βέβαια πολύ ευχάριστο να μαθαίνουμε ότι μπορεί να παραγνωρίσει το Συμβούλιο την γνωμοδότησή μας. Ναι, ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος που σας το είπα. Ε, απλώς θέλω να εξηγήσω τη διαδικασία, κυρία Κρέλ. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι ωραίο όμως να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα θέλαμε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ω κοινοβούλιο, η μόνη ευκαιρία που έχουμε, νομίζω, να εκφράσουμε τη γνώμη μα πρέπει να αξιοποιηθεί. Μια επιστολή, λοιπόν, τη Προέδρου, έστω, πρέπει να υπάρξει, πρέπει να την αξιοποιήσουμε και βεβαίω έχουμε συζητήσει και για τη ζάχαρη αλλά και για την μπανάνα όπω λέγατε. Και φτάσαμε τελικά ε, στο συμπέρασμα ότι οι εξόχω απόκεντρε περιοχέ πρέπει να έχουν μια ειδική μεταχείριση και πρέπει αυτό να το καταστήσουμε σαφέ με μια επιστολή που θα γράψουμε, θα γράψει σε σύντανότα ε, σήμερα. Αλλά θέλω και στην επιστολή αυτή να υπάρξει μια ε, υποσημείωση, μια υπόμνηση ότι θα ε, εντατικοποιήσουμε την επεξεργασία τέτοιου είδους θεμάτων και θα εκφράζουμε πολύ πιο ξεκάθαρα τις θέσεις μας ώστε να μην μπορεί το Συμβούλιο να μας ε, σαρώνει με τέτοιου είδους βραχυπρόθεσμες και πιεστικές αποφάσεις. Ο είναι νομίζω. Ευχαριστώ. Δεν θα σχολιάσω τα διαδικαστικά του Συμβουλίου και την καθυστέρηση του Συμβουλίου. Εγώ θέλω να τονίσω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι πνιγόμαστε μέσα σε ένα ποτήρι νερό αυτή τη στιγμή δεν ε, δημιουργήθηκε τώρα αυτή η κατάσταση. Πρόκειται για συγκεκριμένες διατάξεις της συνθήκης όπου προβλέπεται ότι οι εξόγως απόκεντρες σε περιοχές λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους δικαιούνται θετική διακριτική μεταχείριση σε ορισμένες περιπτώσεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων όπως ε, στην προκειμένη περίπτωση το ρούμι των ε, εξόγως απόκεντρων περιοχών της Γαλλίας και λέμε ότι ενδέχεται να δημιουργήσουν δημιουργήσουν συγγνώμη, στρέβλωση στην εσωτερική αγορά των ε, ινοπνευματοδών, ε, νομίζω είναι παράλογο να ανησυχούμε τώρα με το ρούμι των ε, υπερπόντιων ε, της Γαλλίας και να μην ασχολούμαστε με το Πακιστάν, με τις μπανάνες της Κολομβίας Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν ασχολούμαστε με ουσιαστικά πράγματα και μας απασχολούν ε, λεπτομέρειες ε, ουσιαστικά. Ε, το ΕΛΚ τίποτα δεν έχει καμία ένσταση. Θέλουμε να ακολουθηθεί όπως στο παρελθόν η ίδια διαδικασία, όπως για τα, τις Κανάριες νήσους. Απλουστευμένη λοιπόν η διαδικασία του Άρτς 46. Αυτά. Ευχαριστώ Γιούνους μαζί. Ναι, ε, προφανέστατα είμαστε υπέρ της ε, απλουστευμένης διαδικασίας. Ε, δεν θα υψέλθω σε λεπτομέρειες. Είναι και χρονικό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό να εγκριθεί στις αρχές του χρόνου η πρόταση από την Ολομέλη. Εξάλλου θεωρώ ότι ε, είναι θεμητό από πλευρά του Κοινοβουλίου να ε, εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση, την καθυστερημένη υποβολή της αίτησης από πλευρά του Συμβουλίου. Σήμερα το πρωί συζητούσαμε το θέμα των ε, από κέντρων περιοχών και το, την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερη κατάσταση που επικρατεί σε αυτές τις περιοχές ε, από πλευράς Επιτροπής και της Ένωσης λόγω της μεγάλης απόστασης ε, των που χωρίζουν τις αγορές αυτών των περιοχών από την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ε, το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα υπερπόντια εδάφη δεν νομίζω να δημιουργεί πρόβλημα σε κανέναν. τάχιστα θέλουμε να εγκριθεί ιδέα από την Ολομέλεια, οπότε δίνουμε τη συγκατάθεσή μας ώστε να μπορέσετε να προσφύγετε στο το, στη διαδικασία άρθρου 46. σε ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα και ο Γέννης έχει ζητήσει το λόγο. Θέλεις να μιλήσεις Γεννη. Όχι, δεν θέλεις. Η Μαρή Τερέζ έχει ζητήσει το λόγο. Ναι, πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως με τον Όνο Τεσέιρα και τον ε, ε Μαρζή. Ε, καλά δεν είναι και τίποτα, δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Δεν κάνουμε έτσι, πρώτο αυτό. Και δεύτερον, ε, όλοι γνωρίζουμε τι ιδιαιτερότητε των και απόκεντρων περιοχών, τι ιδιαιτερότητε από οικονομική πλευρά, από πλευρά απόσταση, και άρα νομίζω θα έπρεπε να υποστηρίξουμε αυτή την προσέγγιση παρότι όντως πρέπει να καταγγείλουμε την καθυστέρηση που σημειώνεται από πλευρά του Συμβουλίου. Αύριο όταν κληθούμε να εγκρίνουμε τις προτάσεις εγώ προσωπικά θα τις υποστηρίξω. Ευχαριστούμε Νίκολσον. Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ 100% με τόσο η κυρία Μπέρντερ τελικά προσπαθούμε να διευκολύνουμε τις ε, εξόχους απόγεντες περιοχές. Υπάρχει όμως, είναι γεγονός ότι υπάρχει εδώ πέρα στρέβλωση της αγοράς και αυτό θα συνεχιστεί 7 χρόνια στο μέλλον. Εντάξει, τότε αν αποφασίσουμε ότι δεν μας νοιάζει η ενιαία αγορά, καλώς. Αλλά είναι λάθος το ότι τόσο αργά το Συμβούλιο κατέληξε εκεί που κατέληξε. Είναι επίσης λάθος 100% το ότι ανεχόμαστε το Συμβούλιο το οποίο κάνει ό,τι θέλει και αγνοούν το Κοινοβούλιο. Όχι, να ακολουθήσουμε την συνήθη τακτική διαδικασία και όχι την συντομευμένη. Δεν φταίει η δική μας Επιτροπή για αυτά τα οποία έγιναν. Προσπα... Επίσης, ε, εάν ακολουθηθεί η συντομευμένη διαδικασία, τότε δημιουργούμε προηγούμενο για το μέλλον Οπότε μπορεί να ξαναγίνουν τα ίδια. Άλβες. Ευχαριστώ. Θέλω να τονίσω μία μόνο διάσταση του ζητήματος, ε, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο θα πρέπει ε, να κάνει εμπρόθεσμα τις προτάσεις του και δεν θεωρώ ε, ότι πρέπει να επαναλαμβάνεται διαρκώς αυτό διότι γνωρίζει πολύ νωρίτερα τις προθεσμίες που πρέπει να τηρήσει. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα το να τα μπλέκουμε όλα μεταξύ τους, δηλαδή ε, έχουμε ε, από μακρισμένες περιοχές, εκατοντάδες χιλιόμετρα απέχουν από την εσωτερική αγορά και τι λέμε, έχουμε παρανοήσει, μου φαίνεται εντελώς παράλογο να μιλάμε γι' αυτό το ζήτημα. Ε, στο ε, ε, ξέρουμε όλοι τι γινόταν στο Σουρινάμι και στην Γουινέα παραδείγματο χάρη πηγαίνανε, μπαίνανε στα σκαφάκια τα μικρά οι άνθρωποι και πηγαίνανε από την άλλη πλευρά για να κάνουν τα ψώνια του. Εμεί δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε αυτό. Υπάρχει ούτως ή άλλως εξωτερικός ανταγωνισμός και από αυτό πάσχουμε όχι από τη στρέβλωση που μπορεί να δημιουργήσει αυτή η λιγοστή εξωτερικος ανταγωνισμος και ποσότητα ε, ε, προϊόντων που προέρχονται από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές ε, της Ένωσης. Ε, πρόεδρος, ευχαριστώ. Η λιγοστη ποσοτητα προιοντων που προερχονται απο τι εξοχω αποκεντρε περιοχέ τη Ένωση ε ευχαριστω η επιτροπη Επιτροπή. Ε, υπάρχει κάποιος εκπρόσωπός της θα ήθελε να πάρει το λόγο για αυτό το ζήτημα. Ε, συμβούλιο, οποιοδήποτε τέλο πάντων. Ναι κύριε Πρόεδρε, κάποια γενικόλογο θα σα πω και κατόπιν να δώσετε στον συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με τα ε, τελωνιακά, φορολογικά υπάρχουν μειωμένοι εμείς κατανάλωση κατανάλωσης ε, σύμφωνα με το άρθρο 349 τη συνθήκη και, και αυτό προβλέπεται για τα υπερποντιά δάχτυλα και οπότε ε, υπάρχει αυτή η πρόβλεψη ακριβώ γιατί λαμβάνεται υπόψη το πόσο απόμακρυνες αυτέ τι περιοχέ, ότι είναι νησιωτικέ ε, κλπ. κλπ. Και αυτό προβλέπεται για κάποιο μικρό αριθμό προϊόντων. Οπότε έχουμε αυτή τη διάταξη τη συνθήκη που ακριβώς ε, προβλέπει και διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, οπότε είναι μια σωστή βάση ούτω ώστε να ξεπεραστούν, να αντισταθμιστούν τα, τα, τα, οι έξτρα δαπάνε, το έξτρα κόστο που έχουν να οι επιχειρήσει των περιοχών αυτών. Και οπότε έχουμε την ε, λογοπρόταση πρόταση που ε, έγινε κατόπιν ε, της ε, πρωτοβουλίας της Γαλλίας να παράσει αυτή την προστασία, αυτή την δική μεταχείριση στο Ρούμι που προέρχεται από εκεί για να βοηθήσει τις παραδοσιακές επιχειρήσεις παραγωγού το Ρούμι. Και έτσι να ενισχυθεί η θέση του προϊόντος που παράγεται εκεί. Επομένω, μειωμένο συντελεστή του ΕΜΕΣΟ φόρου κατανάλωση για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστου που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Αν θέλει τώρα μπορεί να συμπληρώσει κάποια στοιχεία ο συνάδελφος από την Γενική Διεύθυνση για φόρους. Επομένως αυτό γίνεται για να αντισταθμιστεί το επιπλέον κόστο, το οποίο φέρουν. Ε, η παραγωγή εκεί, το μισθολογικό επιπλέον κόστος, το πρόβλημα το περιφερμαντικό από την εφαρμογή της κοινωνική νομοθεσίας και κάποια άλλα στοιχεία θέλουμε να καλύψουμε όσον αφορά τη θέση σε εμπορία του Ρουμιού. Ε, οι μπουκάλες είναι πιο μεγάλες και έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Και γι' αυτό και προβλέπονται αυτές οι εξαιρέσεις, οι παρεκκλήσεις ε, με νομική βάση το άρθρο 349 ούτως ώστε να προσαρμοστεί η φορολογική τελωνική νομοθεσία τη ε, κοινότητα, λαμβάνοντα υπόψη τις διορυθμίες, διοτυπίες αυτών των ε, περιφερειών και επομένω λαμβάνεται το 349 το άρθρο που αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ε, εν συνόψη, αυτό είναι το αντικείμενο, ο σκοπός της ε, πρότασής μας. Ελπίζω να απαντήσουμε στην ερώτηση. Δεν ξέρω αν κάποιος ήθελε να υποβάλει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, ο κύριος Νίκολσον. Από ό,τι κατάλαβα. Έχουμε αυτή την ε, παρέκκληση η οποία ισχύει από το 1988. Θα ήθελα να ρωτήσω ε, τον ε, αρμόδιο για τα φορολογικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πότε, εάν κάποτε προβλέπουν την κατάργηση αυτής της παρεξήτη τι, είναι, θα ισχύει ΕΣΑΗ. Ευχαριστώ, δεν θέλει άλλο το λόγο οπότε όχι μπορεί να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Α, μισό εδώ ο κ. Μποστινός το λόγο. Μία ερώτηση μόνο κύριε Πρόεδρε. Είναι δυνατόν με απλά λόγια να πούμε το ότι αποτελεί κάτι σαν οπτάου, σαν αυτοεξαίρεση ε, αυτή, αυτή, αυτή η διάταξη, αυτή η πρόταση για τις, ε, για τις περιφέρειες αυτές. Αυτό προσπαθώ να μας εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος, ότι υπάρχουν αυτά τα δικά προγράμματα για τις εξόχους, εξόχως τις περιφέρειες, για να αντισταθμιστούν κάποια άλλα προβλήματα. Τέλος πάντων, να τους ξαναδώσουμε το λόγο. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις ε, ερωτήσεις. Ξανά έχετε το λόγο. Η μία ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος, ήταν το κατά πόσον πρόκειται για κάποια παρέκκληση που έχει ε, ημερομηνία λήξεως. έχει μόνιμο χαρακτήρα διαρκή δηλαδή ή θεωρείτε ότι δεν θα χρειάζεται, δεν θα χρειάζονται αυτές οι περιφέρειες ε, αυτήν την παρέκκληση. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το μέτρο προβλέπεται να έχει διάρκεια 7 χρόνια. έχει περιφερειακό χαρακτήρα, πρόκειται για κρατική ενίσχυση και προβλέπεται να επανεξετάζεται κάθε 7 χρόνια. Οπότε και για μας αυτό είναι μια ευκαιρία κάθε 7 χρόνια να το μελετούμε. Ε, κοιτάξτε, η, απόσταση που χωρίζει από εμά αυτές τις περιφέρειες δεν θα έχει μειωθεί σε 7 χρόνια. Όμως μπορεί να έχουμε οικονομικές εξελίξεις διαφορετικές. Οπότε γι' αυτό προβλέπεται αυτού του είδους ο χρονικός ε, περιορισμός, αυτού του είδους η χρονική διάρκεια του μέτρου, ούτω ώστε να έχουμε σε τακτά διαστήματα την εξέταση για να αντισταθμίζουμε το μειονέκτημα, το επιπλέον κόστος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι εκεί. Οι δεγαλικές αρχές θα πρέπει ενδιάμεσα να συντάσσουν και να μας υποβάλουν μια έκθεση σε σχέση με το πώς εξελίχθηκε εκεί η κατάσταση, τι γίνεται με τις επιπλέον δαπάνες, αν ανέβηκαν, αν μειώθηκαν και ελπίζουμε να απαντήσαμε η Πρόεδρος. Ναι, για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, θα λάβει το λόγο η Κατρίν Μπέρντερ και ελπίζουμε να είναι η τελευταία που λαμβάνει το λόγο. Ναι, έχω μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, Να μα πούνε μήπω έχουν υπόψη του Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ΠΟΕ για αυτού του είδους τις ε, επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις τέλο πάντων για το προϊόν αυτό. Γιατί όπως είπε ο Τζιμ, πρόκειται για στρέβλωση. 20 χρόνια. Σύμφωνοι, είναι απομακρυσμένες αυτές οι περιφέρειες, αλλά η μεταφορά το μεταφορικά μέσα τέλο πάντων. Τώρα είναι γρηγορότερα. Ε, πόσο πια παίρνει το ρούμι να φτάσει στην επιδοτική ε, Ευρώπη. Είναι τρομερέ ποσότητε ρουμιού που έρχονται και στρεβλώνουν την αγορά στην Γαλλία. Μπορεί να απαντήσει, λέει η πρόεδρο. Σε σχέση με την κοινή πολιτική, σε σχέση με τον ΠΟΕ, εντάξει, ξέρουμε ότι προβλέπεται από ένα άρθρο αυτή η ειδική μεταχείριση. Επιτροπή. Αυτό που μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σα είναι ότι σήμερα δεν προβλέπεται κάποιο ένδικο μέσο όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κάτι σαν προδικαστικό ερώτημα ε, ούτε για το 10 επομένως ούτε και για τον Οργανισμό Εμπορίου τον τίποτε προς το παρόν. Ναι, Λουίς, θα δώσω το λόγο, λες τον κύριο Άλβες, αλλά... Άλβες. Θέλω να υποβάλω στην ε, Κομισιόν μία ερώτηση. Ισχύει αυτός ο κανονισμός εδώ και 7 χρόνια και ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ και πόσα χρόνια απέχουν τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα ε, τι θα γίνει, θα πλησιάσουν γιατί θα πρέπει αυτό το μέτρο να καταργηθεί. Είναι μακριά αυτές οι απόγεντρες. Μήπως θέλετε να ξαναπαντήσετε με τον ίδιο τρόπο. Ξέρω τι να σας πω, έτσι όπως αλλάζει, όπως αλλάζει το κλίμα της γης μπορεί να αλλάξει και η απόσταση. Καλά εντάξει πέραν τώρα των αστείων. Μπορεί να μας αρέσει η εν λόγω διαδικασία, αλλά όπως θα έπρεπε να γνωρίζουν οι Βρετανοί συνάδελφοι, ε, για τα φορολογικά υπάρχει εθνική αρμοδιότητα. Έχουμε εμείς ως Κοινοβούλιο πολύ περιορισμένη αρμοδιότητα γι' αυτό. Έχουμε αυτή την διαβούλευση, έχουμε δικαίωμα γνωμοδότησης. τι να κάνουμε τώρα. Οπότε σας ερωτώ, συμφωνείτε να ακολουθήσουμε την διαδικασία του άρθρου 46. Ε, νομίζω οι βασικές πολιτικές ομάδες ε, αυτό θέλουν. Επίσης, η Κατρίν Μπέρντερ είπε ότι να γίνει μια συζήτηση, αλλά κάτι να γίνει αυτή η συζήτηση στην επόμενη θητεία. Αλλά να μην το ξεχάσουμε το θέμα, να το συζητήσουμε. Και να δούμε τι θα γίνει με τις εξόχως απογοητεύσεις περιφέρειες και αυτή την προτιμησιακή μεταχείριση που επιφυλάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βέβαια αισθάνεται ιδιαίτερη ευθύνη για αυτές τις ε, περιοχές η Ευρώπη. Και εμεί ω Περιφερειακή Επιτροπή θα πρέπει να δούμε τι λύσει μπορούν να δοθούν και να δούμε στο μέλλον τι θα κάνουμε. Άρα, όλοι όσοι ξαναεκλεγούν, να τους θυμίσει, σε όλους τους εκλεγούν τέλος πάντων, να τους θυμίσει η γραμματεία ότι πρέπει αυτό να συζητηθεί. Πάντως, εδώ και τώρα πρέπει να αποφασίσουμε για το κατά πόσο θα συμφωνήσουμε αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία εκείνη που σας πρότεινα. Η διαδικασία του άρθρου 46 ποιοι είναι υπέρ να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Όχι, δεν θέλω να μάθω ποιοι είναι κατά, θέλω να μάθω και ποιοι είναι υπέρ. Θετικά τοποθετηθείτε. Καλά, τώρα ποιοι είναι κατά. We don't have 10. We need 10 to... Α, δεν έχουμε 10 ψήφους. Απαιτούνται 10. What you want to change, but... okay, so we... Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Άρα, προχωρούμε. Επί τη βάση του διαδικασίας 46. και επομένω θα αναλάβω εγώ να ακολουθήσω τη διαδικασία αυτή ω πρόεδρο. Πάει αυτό το σημείο και πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 9 τη μεσή διατάξεω. Ρώσα Σταρά Φεραγκούτ. Ταμείο Αλληλεγγύη. Ρώσα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για αυτή την έκθεση που αφορά το Ταμείο Ελληνική, όπως ξέρετε συγκροτήθηκε το 2002, ούτω ώστε να εκφράσουμε την ευρωπαϊκή ελεγγύη ε, όσον αφορά κάποιες θεομηνίε, κάποιες καταστροφές και ε, όσο ισχύει αυτό το ταμείο, όσο υπάρχει αυτό το ταμείο, εντοπίστηκαν κάποιες δυσκολίε στη λειτουργία του. Επομένω, είπαμε ότι το πιο σωστό είναι να συντάξουμε αυτή την ε, έκθεση που θα προτείνει τρόπους άρσιος αυτών των προβλημάτων. Το ταμείο αυτό αφορά αυτές τις θεομηνίες που έχουν περιφερειακό χαρακτήρα και το 2005 έγινε προσπάθεια ε, αλλαγής, τροποποίησης και είπαμε να γεννηθούμε στο ίδιο πνεύμα αλλά να τροποποιήσουμε όλα όσα δεν θεωρήθηκε ότι είναι αποδοτικά αποτελεσματικά σε σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου. Τώρα, όσον αφορά τις περιφερειακές θεομηνίες και καταστροφές, είπαμε ότι ισχύει ο κανονισμός ε, που προβλέπεται και ενεργοποιεί το Ταμείο. Όποτε σε συγκεκριμένη περιφέρεια πλήσεται η πλειοψηφία του πληθυσμού όσον αφορά τις σοβαρές επιπτώσεις της καταστροφής. Βεβαίως ε, δημιουργούνται προσδοκίες έτσι ε, στις περιφέρειες και επομένως η Επιτροπή των Περιφερειών και η Κομισιόν ε, είπαν ότι θα πρέπει να κινητοποιείται το 1%, η Κομισιόν είπε 1,5% σαν κατόφλι ζημίας. Και είπαμε ότι θα πρέπει για τις σοβαρές καταστροφές να ισχύουν τα ίδια βάσει του ισχύοντος κανονισμού. Όποτε επομένω υπάρχει μια καταστροφή πάνω από το κατόφλι καταστροφής και προβλέπονται τέλο διάφορα ποσά τώρα για αυτό το ε, είπαμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 0,6 του ΑΕΠ ως προκαταβολή θα πρέπει να προβλέπετε κάτι και είπαμε ότι έχουμε ως μάξιμου 30 εκατομμύρια ευρώ είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15% η Επιτροπή των Περιφερειών και λέμε και εμείς και φτάνουμε σε ένα μάξιμου 40 εκατομμύριων επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται το, ταμείο αυτό για τεχνική βοήθεια. Αυτό το έχει προτείνει η Επιτροπή των Περιφερειών μέχρι το 1% του συνόλου το, της του ταμείου το οποίο να αφορά κάποια ανασυγκρότηση των υποδομών αλλά και την κυριτικότητα αυτών των, ε, των υποδομών. Η προθεσμία είναι 10 εβδομάδες. Αίτηση κινητοποίηση. Και εμείς είπαμε να γίνει ε, αυτό το χρονικό διάστημα 15 εβδομάδες για να υπάρχει περισσότερη ευελιξία. Και η εκτέλεση, η υλοποίηση προβλέπεται να είναι ένα έτος. Εμείς προτείναμε 1,5. 18 μήνες. Κάτι άλλο καινούργιο το οποίο τώρα εμείς προτείνουμε είναι να ισχύει αυτό για τις περιοχές 2 και 3. Τις κατηγορίες 2 και 3. Ανάλογα με τον πληθυσμό των περιφερειών αυτών. Θα έχουμε τώρα την ε, Ελληνική Προεδρία, θα συνεργαστούμε με την μόνιμη την γιατί τρέχουν αυτές οι προθεσμίες, τόσο ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τους τριμερείς διαλόγους, να συμφωνήσουμε και συνεργάστηκα και με την Επιτροπή των Περιφερειών γιατί και από εκεί υπήρχαν πάρα πολλά αιτήματα. Έχουμε πολλές προπολογίες να βελτιωθεί το κείμενο. Αλλά να μην αλλοιώσουμε την, ε, το σκοπό του Ταμείου, γιατί από το ενδύσεις περάσαμε στα στο, στο, στο μισό δι, στα 500 εκατομμύρια. Βεβαίω και έχουμε την οικονομική συγκυρία, αλλά θα πρέπει να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που μέχρι σήμερα ε, προέκυψαν, γιατί βεβαίω και έχει δημιουργήσει πολλές προσδοκίες αυτό το ταμείο. Ευχαριστούμε. Παύλ Πράντα από την Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι ο εκεί εισηγητής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά κυρίες και κύριοι βουλευτές για την πρόσκληση στην Επιτροπή των Περιφερειακών Υποθέσεων. Θα ήθελα εκ μέρους της ε, ε, Επιτροπής των Περιφερειών να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς ε, την ε, κυρία συναδέλφο για την πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή μας. Πάντοτε ε, μας ε, έδωσε χρόνο για να συνομιλούμε. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές. Ακούστηκαν λοιπόν εδώ οι προτάσεις και ανταποκρίνονται τα όσα είχαμε συζητήσει Είναι καταγεγραμμένη πρόταση. Ταμείο Ελεγγύης λοιπόν το οποίο ναι είναι κατά κύριο λόγο εγκατεστημένο στα ε, κρατη αλλά ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη σημασία στα, σε τοπικό επίπεδο. Εμείς στην περιοχή μας έχουμε πολύ συχνά πλημμύρες, παραδείγματι. Είμαστε στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχίας και έχουμε αξιοποιήσει πολλές φορές αυτό το ταμείο, το 2010 ε, ήδη και έχουμε αρκετή εμπειρία ε, για το πώς θα θέλαμε να διαμορφωθεί ε, η κατάσταση. Δεν έχω πολλά να προσθέσω όσο είπε η κυρία Στρέλιας. Έχουμε συμφωνήσει στα πιστρεκτων των ζητημάτων. Ένα-δύο μόνο πράγματα που θα μπορούσα να προσθέσω γιατί δεν αντικατοπτρίζονται 100% τα δικά μας μελήματα στην έκθεση. Καταρχάς, ο περιορισμός του κριτηρίου, η μείωση του κριτηρίου του 1,5% στο 1% για την προσβαλλόμενη περιοχή. Νομίζω ότι αντικα το πολύ καλύτερα την ε, κατάσταση, ιδιαίτερα σε περίπτωση περιφερειακού τύπου ε, φυσικών καταστροφών για την υποστήριξη από το Ταμείο. Ταχνικό όμως ε, το ζήτημα πάνω απ' όλα. Και άλλη μία πρόταση στην οποία θα ήθελα να σου την υποστήριξη σας. Θα ήθελα να ληφθεί υπόψη αυτή η ιδιαιτερότητα των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Η ΝΑΤΣ που ε, βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη και αντιστοιχούν σε μια κατηγορία Nats ουσιαστικά, αλλά επειδή βρίσκονται κοντά στα σύνορα είναι είναι 3, νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μία περιφέρεια. Μία περιφέρεια ώστε να εφαρμόζεται, να τηρείται το περιφερειακό κριτήριο σε αυτές όταν πλήττονται από μια φυσική καταστροφή. Νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα πολύ θετικό μήνυμα για τους πολίτες. Δεν βλέπουμε πάντα κάθε θητεία του Κοινοβουλίου και σε κάθε πολιτική να προσθέτει ε, κάτι το θετικό στις πολιτικές μας, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω μπορούμε να έχουμε μια πραγματική προσθέμενη αξία ανταποκρινόμενη στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Και γι' αυτό παρακαλώ να λάβετε υπόψη και να δεχθείτε αυτή την πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών. Έχουμε την εμπειρία με στις περιοχές μας. Αν ε, ε, έχουμε πλημμύρες στην Τσεχία, μέσα σε λίγες ώρες τα, ε, η πλημμύρια θα πλήξει και την Πολωνία και τη ε, Γερμανία επίσης. Είναι κάτι το οποίο δεν ελέγχεται μέσα εθνικά σύνορα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μιλάμε για περιφέρειες. Και το πιο σημαντικό μας αίτημα είναι αυτό. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να το λάβετε υπόψη. Και πάντα ε, ευχαριστώ, όπως είπα, για την πολύ καλή συνεργασία μέχρι τώρα. Είμαστε σε οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Η ε, Κριστίν Βεστφάλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Ταμείο Ελεγγύης είναι για μένα το πιο σημαντικό εργαλείο που μπορεί στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και μάλιστα γρήγορα. Πιστεύω επίσης ότι πρόκειται για ένα μέσο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιδείξει την αλληλεγγύη της με τις ε, πληττόμενες περιοχές. Ε, και γι' αυτό νομίζω ότι και πέραν των δερφωτικών ταμείων που έχουμε ήδη συζητήσει και που ολοκληρώσαμε πλέον, ε, δείχνει το Ταμείο αυτό αλληλεγγύη στους πολίτες πόσο ξεκάθαρη βοήθεια μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όπως με τις ε, πλημμύρες και το 2012 η Αυστρία, η Γερμανία, η Τσεχία μπόρεσαν, γιατί και εγώ από μια τέτοια περιοχή που επλήγει από τις καταστροφές ε, προέρχομαι μπόρεσαν λοιπόν να ωφεληθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης και νομίζω ότι θα πρέπει όπως πρότεινε οι συνάδελφες αλλά και εσείς από, το, από την Επιτροπή των Περιφερειών να, αξιοποιηθεί, το Ταμείο. Πολύ συχνά όμως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι πολύ κοπιαστικές και βαριές, κρατούν Πολλοί οι προθεσμίες για τη διάθεση των κονδυλίων. Οι περιοχές αυτές περιεμένουν ε, ε, επιματέω για την ε, καταβολή των κονδυλίων όταν κατάει πάρα πολύ αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία η οποία θα έπρεπε κανονικά να είναι πολύ πιο απλή και να προσφέρονται ταχύτατα οι ενισχύσεις, η βοήθεια στις περιοχές αυτές των έχουν πληγεί. Ε, ενδιαφέρον είναι να έχουμε σαφείς ορισμούς, ενδιαφέρον είναι επίσης να έχουμε απλή διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων. Αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα, αλλά επίσης και η ιδέα μιας προκαταβολής αποζημιώσεως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το σχέδιο εκθέσεως της συναδέλφου που έχει κατευθεί και για μετάφραση από την Παρασκευή ε, νομίζω ότι ορίζει πάρα πολύ σημαντικά ορόσημα ε, δεν έχω πάρα πολλά να προσθέσω στα όσα είπαν οι συνάδελφός μας αλλά και ο κύριος από, το από την Επιτροπή των Περιφερειών. Πρέπει λοιπόν ε, να τα δεχθούμε όλα αυτά και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι προβλέπεται για τον Ιανουάριο μια ακρόαση για το Ταμείο Ηλεγγύης γιατί έτσι μπορούμε πιστεύω στην ουσία να συναντήσουμε τους ανθρώπους από τις, πληγόμενες, ε, τις πλησόμενες περιοχές, δημάρχους και το καθεξής εκπροσώπους των πολιτών για να δούμε τι είδους αιτήματα ζητήματα έχουν να εκφράσουν και τι άλλο θα πρέπει να αλλάξει στο Ταμείο Αυτό Αλληλεγγύης. Θα μας απασχολήσει λοιπόν και στο μέλλον. Και επίσης ε, πέραν της ακροάσεως για την οποία αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω και για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ, Και Ο Νίκος, παρακαλώ. Όχι, κυρία Σρέτερ, Ελίζα Μπέτες, εκπροσωπής Ναι, εκπροσωπώ τον Νίκο Χουντή. Χρυσόγγελο, συγγνώμη, ο οποίο έχει ασχοληθεί βέβαια με το θέμα αυτό και ω Έλληνα έχει συχνά να αντιμετωπίσει του είδου φυσικέ καταστροφέ. Πολλέ είναι οι περιοχέ οι οποίε μένουν πολλέ φορέ αφανεί, όπω η παραδείγματι στην ε, Ρουμανία και τι μεγάλε καταστροφέ στην περιοχή των Καρπαθίων είτε πρόκειται για πλημμύρες, είτε πρόκειται για νεροποντές, ε, υπάρχει ανάγκη για άμεση βοήθεια. Θυμάμαι επίσης πάρα πολύ καλά ότι ο Επίτροπος Μπαρνιέ σε μια περίπτωση όπου είχαν πληγεί από πλημμύρες πάρα πολλές περιοχές το 2002 ήταν και στη Δρέσδη την διατηρή μου πατρίδα όπου ξεκάθαρα είχε δηλώσει ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό μέτρο. Θυμάμαι πολύ καλά την ε, ομιλία του, στην οποία είχε χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τον όρο ε, πρόληψη και βέβαια το Κοινοβούλιο επικρότησε. Πρώτη τοποθέτηση αυτή, από εκεί και μετά ο κύριος Μπαρνιέ και όσο ήταν επίτροπος για τα περιφερειακά δραστηριοποιήθηκε για να αναπτύξει αυτό το μέτρο, αυτό το μέσον στην διάσταση της πρόληψης ιδιαίτερος με τις επενδύσεις που χρειάζονται ώστε να μην χρειάζεται μόνο να διορθώνουμε τη ζημιά αλλά να βλέπουμε και να αναλογιζόμαστε κάθε φορά προκύπτει ένα πρόβλημα τι άλλο πρέπει να αλλάξει για να το αποφύγουμε στο μέλλον γιατί ξέρουμε τι είδους τραγικές συνέπειες μπορούν να έχουν αυτές οι φυσικές καταστροφές για τους εμπλεκόμενους πολίτες. Ιδιαίτερα λοιπόν θέλω να επισημάνω ότι η, υπάρχει ένα, η διαγραφή, η πρόταση για διαγραφή είναι πάρα πολύ εσφαλμένη και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορεί να με το χέρι μας για να το διατηρήσουμε το κομμάτι αυτό. Ο κύριος Άλβες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο Φεραγκούτ και ήθελα να πω ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, δημιουργήθηκε το 2002 για να αντιμετωπίσουμε μεγάλες φυσικές ε, καταστροφές που πλήττουν τα κράτη-μέλη και τις περιοχές μας ε, με ένα επίπεδο ζημιών που απαιτεί επίδειξη αλληλεγγύης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πληθυσμοί βιώνουν δύσκολες στιγμές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανατροπής των οικονομικών δραστηριοτήτων, των πόλεων και των περιοχών και εκεί βλέπουμε ότι σε τέτοιες στιγμές ε, είναι που χρειάζονται οι πολίτες τη βοήθεια και την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα αντίδραση του το Ταμείου, την ε, δυναμικότητά του να επέμβει σε αυτές τις περιοχές, εισαγάγοντας την έννοια της περιφερειακής φυσικής καταστροφής. Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στα συγκεκριμένα προβλήματα των επιμέρους περιοχών. Είδαμε από το 2002 όταν δημιουργήθηκε το Ταμείο ότι το, η εστίαση ήταν στις ε, εξόχους απόκεντρες περιοχές ε, βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού. Τώρα όμως ε, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι πλέον ευάλωτες περιοχές ως προς τους κατακλυσμούς και τις φυσικές καταστροφές και θεομηνίες. Διαπιστώνουμε επίσης ότι οι νησιωτικές περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα αλλά όμως δεν φτάνουν το ποσοστό του ΑΕΠ που χρησιμοποιείται ως κριτήριο για την επέμβαση του Ταμείου, ώστε να μπορέσουν να συνεχιστούν οι ε, συνηθισμένες οικονομικές δραστηριότητες. Και βλέπουμε λοιπόν ότι πλήττονται βασικοί τομείς της οικονομίας ή βασικές υποδομές όπως οι δρόμοι, οι δικές αρτηρίες και οι λιμένες. Χρειάζεται προσαρμογή στις ιδιαίτερες καταστάσεις λοιπόν. Δεν μπορούμε να έχουμε ενιαίο ποσοστό 1,5% του ΑΕΠ θα πρέπει να μειωθεί στο 1% ούτως ώστε η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στο μέτρο των αναγκών των ε, πλέον ευπαθών περιοχών των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει επίσης να έχουμε την δυνατότητα όταν χρειάζεται να προβλέψουμε εκτοπισμό των υποδομών που έχουν πληγεί ούτως ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά πλήγματα από φυσικές καταστροφές όταν διαπιστώνουμε ότι επανειλημμένα πλήττεται μία υποδομή ή μία περιοχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης μπορεί να λειτουργεί εδώ και λίγο διάστημα, αλλά έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα και θα ήθελα να ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία. Έλαβε υπόψη πολλές ε, πραγματικές καταστάσεις στην έκθεσή της και βλέπω ότι λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που έχουμε γνωρίσει σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης. Ε, έτσι λοιπόν και με την ε, δυνατότητα αυτή που δόθηκε για συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή ε, έκθεση. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή να προχωρήσουμε παράλληλα με την Επιτροπή των Περιφερειών και πιστεύω ότι ιδιαίτερα οι δήμαρχοι των περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές μπορούν να μας ε, ε, στηρίξουν, να μας προσφέρουν τη βοήθειά τους για πιο καλή ακόμη δουλειά. Ένα-δύο ζητήματα θα ήθελα να επισημάνω που θα ήταν σκόπιμο να μπουν πιστεύω στο κείμενο. Καταρχάς τη δυνατότητα η πληττόμενες υποδομές να προστατευτούν μεταφερόμενες σε άλλες περιοχές όπου δεν υπάρχουν προβλήματα. Ε, και έτσι θα πρέπει να υπάρχει ένας χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης η προθεσμία για την ε, προσφορά των ε, υπηρεσιών της ενίσχυσης δεν θα πρέπει να καθυστερεί. Πρέπει το ταχύτερο δυνατό να προσφέρεται αυτή η ενίσχυση. Η προκαταβολή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και πάλι Κλείνοντας, ευχαριστώ τους δύο συναδέλφους, την κυρία εισηγήτρια, αλλά και τον κύριο Μπράντερ από την Επιτροπή των Περιφερειών και ελπίζω να συνεχιστεί με έτσι καλή συνεργασία και στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριο Μποστινάρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, χαιρετίζω την έκθεση και τονίζω τη σημασία της. Ε, θα ήθελα να πω ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη συνάδελφο που επέστρεψε την προσοχή μου στην σημασία αυτού του ζητήματος. Λοιπόν, τρεις είναι βασικές συνιστότησες. Πρώτα απ' όλα η πρόληψη, ε, όταν μιλάμε για φυσικές καταστροφές, ε, πλημμύρες, σεισμούς, είτε μιλάμε για άλλες θεομηνίες Το γεγονός είναι ότι ε, κατά την εκπόνηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης τονίσαμε τη σημασία εκπόνησης προγραμμάτων ε, οικοδόμησης υποδομών που ε, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τις φυσικές καταστροφές. Χρειαζόμαστε περιφερειακά ή διαπεριφερειακά κέντρα, τα οποία ε, θα μας επιτρέπουν εξοικονόμηση πόρων μέσω μιας αποτελεσματικής, ε, ευέλικτης ευέλικτης χρήσης τους ανεξαρτήτως εκτός της ε, γεωγραφικής θέσης όπου σημειώνεται η φυσική καταστροφή. Δηλαδή ε, θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση αυτά τα περιφερειακά κέντρα και να επεμβαίνουν όταν ε, συντρέχει λόγος. Όταν δεν επιμένουμε αρκετά στην πρόληψη, τότε απλώς αυξάνονται οι ζημιές σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Δεύτερον, ε, η υλικοτεχνική στήριξη και η χρηστή διαχείριση των πόρων που διαθέτουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό έγκαιρη αντίδραση σε περίπτωση καταστροφών, τουλάχιστον στην περίπτωση πλημμύρα. Είναι απαραίτητο στην υδρογραφική λεκάνη να έχουμε ένα τέτοιο περιφερειακό κέντρο στη Γερμανία, στην Τσεχία, στην Πολωνία, παραδείγματο χάρη, στα σύνορα αυτών των τριών ε, χωρών. Ε, το ίδιο ε, ε, κέντρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την Ουγγαρία και για την Σλοβενία και για τη Ρουμανία. Ξαναλέω, να επικεντρώσουμε την δημιουργία αυτών των κέντρων, μάλλον να βασίσουμε τη δημιουργία αυτών των κέντρων σε κριτήρια όπως υδρογραφικές λεκάνες για τις πλημμύρες συγκεκριμένα. Εάν δεν τονίσουμε παρκώς το σκέλος της πρόληψης και επεμβαίνουμε μόνο εκ των υστέρων ε, μετά την φυσική καταστροφή, ε, θα πολλαπλασιάζονται οι ζημιές. Ε, λόγω των κλιματικών αλλαγών και των ακραίων καιρικών φαινομένων βλέπουμε ότι οι πλημμύρες έχουν καταστροφικά αποτελέσματα στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία σε χώρες ιδιαίτερα αναπτυγμένες με ικανότητες ε, ε, επέμβασης, ε, κρατικές δυνατότητες επέμβασης ζηλευτές, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρκούς αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών λόγω του εύρους τους, των κλιματικών αλλαγών και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή Χρειάζεται μια πραγματική στρατηγική, ούτως και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα κομμάτι της συνολικής μας απάντησης ε, ως προς τα νέα αυτά δεδομένα. Χρειάζεται επίσης ορθότερη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων ώστε να δημιουργήσουμε ένα ε, σωστό πλαίσιο συντονισμού και διαχείρισης ξαναλέω της υλικοτεχνικής υποστήριξης ε, το, ε, μιλάμε για την Ισπανία, για την Ελλάδα για πάρα πολλές χώρες διαπιστώνουμε ότι Πάσχουν οι τοπικές αρχές ε, διότι ε, χρειάζεται ταχύτατη απάντηση σε πολύ ε, ευρεία γεωγραφική ζώνη και δεν επαρκούν οι εθνικές ικανότητες εξού και η ανάγκη ίδρυσης περιφερειακών κέντρων. Χρειαζόμαστε επίσης νέες στρατηγικές με τρόπο να εξασφαλίσουμε συντονισμό όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και διακρατικό συντονισμό και κυρίως διαπεριφερειακό συντονισμό σε επίπεδο υδρογραφικής λεκάνης όπως σας έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, κλείνοντας, ε, ήθελα να πω ότι... στην περίπτωση σεισμών, γιατί ε, ε, μας αυτό μας πλήττει συνήθως στην περιοχή μου, το ίδιο και στη Ρουμανία, στην Ιβυρική Χερσόνησο αλλά και στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην περίπτωση των σεισμών χρειαζόμαστε στρατηγικό σχεδιασμό ε, για να προβλέπουμε τις πιθανές επιπτώσεις όταν σημειώνεται μια τέτοια φυσική καταστροφή ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την απώλεια ανθρωπίνων ζώων και ζημιών φυσικά. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο στρατηγικός ε, σχεδιασμός για να υπάρχει αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Ε, σας συγχαίρω και πάλι για την έκθεση και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, έχουμε μακρύτατο κατάλογο μιλητών. Δεν μπορούμε να υπερβαίνουμε τα 6-7 λεπτά ακόμη, γιατί έχουμε και την Επιτροπή, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Σας παρακαλώ, σύντομα, νου το σέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τάμε θα είμαι σύντομο ε, για... επειδή μα το ζητήσατε. Λοιπόν, ε, συγχαίρω την εισηγήτρια. Ε, πολύ καλή η δουλειά που έκανε και είναι καλή η βάση για τις μελλοντικέ μα εργασίες και για όλες τι τροπολογίες που πρέπει να εισαγαγούμε στο σχέδιο. Ε, συμφωνώ με τον συνάδελφο Ντοσπαλόφ, συμφωνώ σε επιτοπλίστων μαζί του. θα τονίσω μόνο ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Ε, από το 2005 τουλάχιστον μας απασχολεί αυτό το ζήτημα και έχουμε φτάσει στο 2013 και τι έχει συμβεί. Αντίθετα με αυτά που μας είπαν σήμερα κάποιοι συναδελφοί, το Ταμείο Αλληλεγγύης που υποτίθεται ότι είναι ένα εργαλείο ε, ταχείας και αλληλέγγυης επέμβασης, ένα όργανο για να δείξουμε ότι μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους πολίτες. Το αντίθετο έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η βασική πρόκληση στην οποία πρέπει να αντεπεξέλθουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε ε, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής σε τρίτη χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ταχύτατα, σχεδόν στιγμιαία να επεμβαίνει ε, και ιδιαίτερα αλληλέγγυα. Όταν όμως η ίδια φυσική καταστροφή ε, συμβαίνει στο σπίτι μας, σημειώνονται τόσο μεγάλες καθυστερήσει. Ε, λοιπόν, στη Μαδέιρα, στη δική μου περιοχή, δίσε σημειώθηκε φυσική καταστροφή. Πρώτα 2010 ταξινομήθηκε ως μεγάλη φυσική καταστροφή, δηλαδή ε, είχε το, το, κάλυπτε το κριτήριο το 16% του εθνικού ΑΕΠ, ε, ένα δισεκατομμύριο ζημιές ε, λόγω ακραίου καιρικού φαινομένου και σε 16 ώρες συνέβη αυτό. Μέσα σε αυτές τις 16 χώρες καταστράφηκαν 7 χρόνια ε, πολιτικής συνοχής και ακυρώθηκε το ποσό που είχε λάβει η Μαδέιρα μέσω των διαρθρωτικών ταμείων που ήταν ε, το μισό από αυτό των ζημιών. Λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι δεν λειτουργεί σωστά το Ταμείο Αλληλεγγύης και δεν είναι ταχεία η επέμβαση όπως θα έπρεπε. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει με σοβαρότητα ε, να αντιμετωπίσουμε ε, με ειλικρίνεια το πρόβλημα, ούτως ώστε μελλοντικά να μπορούμε τουλάχιστον να επεμβαίνουμε ε, ταχύτατα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε, Κάρενμπαχ. Ευχαριστώ πολύ και πολλά από αυτά που ήθελα να υπογραμμίσω εγώ τα ήδη ο Βίκτορ Ποστινάρου Νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχει το Ταμείο Αυτό Εγώ σε Αυστριακή μπορώ να πω ότι και στην προηγούμενη συνεδρίαση στο Στρασβούργο είχαμε την ευκαιρία να διαθέσουμε 21,6 εκατομμύρια ευρώ για ε, την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πλημμύρες στην Αυστρία από το Ταμείο Αυτό. Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει πάντα να υπογραμμίζουμε είναι ο λόγος για τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης. Είναι στόχος του να καλύψει ζημιές μη προβλέψιμες και ιδιωτικές ακόμη είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε πολύ ξεκάθαρα διότι δεν είναι πάντα αντιληπτό στην Αυστρία. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με ζημιές οι οποίες είναι μη προβλέψιμες και ταυτόχρονα νομίζω θα πρέπει μαζί με την οδηγία για τις ε, πλημμύρες να προχωρήσουμε στην ε, ε, καταγραφή σχεδίων διαχείρισης, στην κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης, τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προβλέψει τι είδου μέτρα προληπτικά πάνω απ' όλα χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις πλημμύρες. Και αυτό όχι μεταθέτοντας την πλημμύρα ε, που εμφανιζόταν σε ένα μέρος της Ευρώπης σε κάποιο άλλο μέρος, αλλά αντιμετωπίζοντας ουσιαστικά το φαινόμενο αυτό. Και όπως υπόθηκε και νωρίτερα, πολύ μεγάλη σημασία έχει για τα προληπτικά μέτρα να διατίθενται τα διαρθρωτικά ταμεία σε συνεργασία με τη χωροταξία, με τη γεωργία, ενδεχομένως μια διαφορετική σύλληψη και αντίληψη για τη γεωργία, γιατί υπάρχουν μεθοδοί παραγωγής οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την δυνατότητα των εδαφών να συγκρατούν τα ύδατα των βροχοπτώσεων. Ξέρετε, στα γερμανικά λέμε όποιο προσφέρει γρήγορα βοήθεια προσφέρει διπλή βοήθεια. Ε, αυτό νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Να είναι μη γραφειοκρατικό αυτό το ταμείο και να προσφέρει το χύτερο δυνατό την βοήθειά του στι πληγήσει περιοχέ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σεκουράκη. Ευχαριστώ πολύ αναγκαστικά ένα τέτοιο θέμα αναδεικνύει πολλά σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν γύρω από το θέμα της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Ε, θα ήθελα και εγώ να εστιάσω κυρίως στο ζήτημα της πρόληψης ε, και να σημειώσω ότι στην Ελλάδα, μιας και γίνεται λόγος και για τέτοιες χώρες, ε, έχουμε τριών ειδών προβλημάτων. Το ένα ζήτημα είναι οι σεισμοί όπως υπόθηκε κιόλας, πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Έχω τη γνώμη ότι πολύ μεγάλο μέρος των, των καταστροφών πρέπει να αντιμετωπίζεται στην φάση της πρόληψης. Εκ των υστέρων τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές είναι ανεπανόρθωτα και πρέπει νομίζω και η έκθεση και γενικά η δράση μας να δώσει πολύ μεγάλη βάση στα ζητήματα της πρόληψης. Μπορώ να σας πω για το παράδειγμα της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη, όπου ορισμένα στοιχειώδη μέτρα αντισυσμικής προστασίας ε, είχαν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, οι καταστροφές ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι σε προηγούμενες δεκαετίες. Όμως, όμως το θέμα της αντισυσμικής προστασίας είναι πάρα πολύ σοβαρό και είμαστε, ε, έχουν γίνει ελάχιστα, ειδικά όσον αφορά την στήριξη ε, δημοσίων κτηρίων, διότι, διότι καταλαβαίνετε αν γίνουν σεισμοί και μετά τρέχουμε να αποζημιώσουμε για ζημιές για τα θύματα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Το ίδιο θέμα αφορά και τις πλημμύρες. Βέβαια, ε, τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες πλημμύρες στη Δυτική Ευρώπη δείξαν ότι κατά τη γνώμη μου είναι αναγκαίες πολύ, σημαντικά έργα υποδομής τα οποία δεν υπήρχαν ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι σε θέση υποδομές που υπάρχουν και στη Δυτική Ευρώπη να αντιμετωπίσουν νέα φαινόμενα. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με εκατοντάδες χιλιόμετρα ε, ρέματα τα οποία έχουν εμπαζωθεί, ρέματα ποταμών δηλαδή, έχουν χτιστεί κτίρια εκεί και κάθε φορά που υπάρχει μια βροχή, μικρή ή μεγάλη, βεβαίως ε, πλημμυρίζει το σύμπαν. Ε, υπάρχει ένα θέμα. Ε, δεν υπάρχει καμία στρατηγική αντιμετώπιση αυτών των μπαζωμένων ρεμάτων. Να ανοίξουν ξανά, να, να μπορούν τα, δηλαδή, τα ποτάμια να βρίσκουν την ε, φυσική τους ε, κήτη και τέτοια προγράμματα δεν υπάρχουν ούτε στο Ταμείο Συνοχής, όπως δεν υπάρχουν ούτε για την σεισμική προστασία. Γι' αυτό και κάθε φορά που γίνεται λόγος για το Ταμείο Συνοχής με ακούτε να, να κάνω κριτική στο ζήτημα αυτό. Τέλος, πυρασφάλεια. Ε, τεράστιο πρόβλημα σε όλο τον Νότο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Μεγάλο πρόβλημα εδώ και το γεγονός ότι υπάρχει μια άναρχη ε, πολιτική ε, οικοδόμηση στα δάση. Μεγάλο πρόβλημα εδώ γιατί υπάρχει μια πολιτική ε, ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης των δασών και των ορεινών όγκων και όσο καιρό υπάρχει αυτή η υπόθεση όσο ταμεία αλληλεγγύης να κάνουμε καταστροφές θα είναι μεγάλες και ακόμα πιο μεγάλες και επίσης δεν υπάρχουν και στοιχειώδη μέτρα πυρασφάλισης, δηλαδή ζώνες αντιπροστα... Ε, ε, πυρηνικής αντιπροστασίας ε, κτλ. κτλ. Και εδώ πάλι από ό,τι βλέπετε υπάρχουν ζητήματα υποδομών. Σε σχέση με αυτό όμως θα ήθελα να σημειώσω ότι σε μια διαδικασία αποψήλωσης της πυροσβεστικής και άλλων σημαντικών δημοσίων υπηρεσιών οι ζημιές είναι επίσης τεράστιες. Α πούμε στην Ελλάδα τα μισά αεροπλάνα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί λόγω τη πολιτική λιτότητα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα, η Κομισιόν και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Οπότε ό,τι και να λέμε το πρόβλημα οξύνεται. Τέλο, ε, νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο το θέμα του ποσοστού των αποζημιώσεων. Κοιτάξτε, πριν δύο χρόνια γίνανε δύο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα έλεγε κανείς ενδεχομένως μικρές πυρκαγιές. Μία στο νησί της Χίου και μία άλλη στην ε, περιοχή της Βιάνου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο νότιο μέρος στην Κρήτη. Στη Μέν Χίο καταστράφηκε όλη η παραγωγή ε, μαστίχας. Ξέρετε, οι άνθρωποι ζουν μόνο από τη μαστίχα, είναι αυτό το ποτό που ξέρετε το ούζο κτλ. Καταστράφηκε η παραγωγή διότι υπήρχε μια πυρκαγιά. Επειδή ήταν χαμηλό το ποσοστό δεν πήραν αποζημίωση. Διότι λέει δεν ανταποκρινόταν στα κριτήρια του ποσού. Στη Βιάνο, στο χωριό από όπου προέρχομαι, καταστράφηκαν σε μία μέρα 120.000 ελιές. 120.000 ελιές. Γίνανε στάχτη. Επίσης δεν πήρανε τίποτα με το επιχείρημα ότι δεν καταστράφηκαν σημαντικές υποδομές που έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ταμείο Συνοχής με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχει μια τραγική κατάσταση ειδικά στο θέμα της ελιάς όπου δεκάδες χιλιάδες οικογένειες για έξι χρόνια δεν έχουν τίποτα γιατί τόσο κάνει το να ε, ε, επανέλθει η παραγωγή. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε θέμα πρόληψης οπωσδήποτε, αλλά υπάρχει και ένα θέμα με το ποσό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Thank you. I would like to ask uh, the Commission... Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο. Σύνομα παρακαλώ, γιατί πρέπει να δευτερολογήσουν οι εσείς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια της Επιτροπής σας γιατί γενικά ε, μας στήριξε στην προσπάθειά μας του Ταμείου Ελληνική και στο έργο μας. Αλλά να σχολιάσω κάποια συγκεκριμένα σημεία και προτάσεις που σήμερα αναφέρθηκαν και που επίσης ε, περιέχονται στην ε, έκθεση. Ξεκινώ από το τελευταίο το οποίο αναφέρθηκε, αλλά το είπαν πολλοί από τους αγορητές. Πρόληψη. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει και ούτε βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Πιο αποτελεσματική είναι η πρόληψη από το, την εκ των υστέρων επέμβαση. Πρόσφατα αναπτύξαμε τέτοιου είδους πολιτική πρόληψης. Ο μηχανισμός ε, πολιτικής προστασίας ε, για τις μέτρα για τις πλημμύρες και με τα μέτρα της συνοχής που ίσχυσαν την περίοδο που τώρα κλείνει είχαμε πάνω από 7 δις για προληπτικά μέτρα. Επίσης, με τη νέα περίοδο χρηματοδότηση θα έχουμε και άλλα δις τα οποία θα επενδυθούν σε FEE e μέτρα πρόληψης. Δεν το ότι ένα ευρώ τη πρόληψη αντιστοιχεί σε πέντε ευρώ το οποίο κανείς θα πρέπει να δαπανίσει για την εκ των υστέρων παρέμβαση. Όλα αυτά όμω πάρα πολύ σημαντικά. Και επίσης δεν θα πρέπει να ανεβάζουμε τον πύχη των προσδοκιών για το Ταμείο ε, Αλληλεγγύης. Φτιάχτηκε το Ταμείο για να καλύψει τις καταστροφές που χτυπάνε παρά τα μέτρα πρόληψη. Γιατί συνεχίζονται φυσικά και οι θεομηνίες και οι καταστροφές, ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος για να αποφύγει τα αυτά τα φαινόμενα. Και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε με τα πεπερασμένα χρηματικά μέσα από τη διάθεσή μας. Έχουμε τις, ε, ε ό,τι προβλέπει το πολιτέ πλαίσιο, το χρηματοδοτικό, και πήγαμε στα 500 εκατομμύρια ετησίω από το 1 δι. Άρα έχουμε αυτού του πόρου, του περιορισμού στη διάθεσή μα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυσκολία το ότι οποιαδήποτε πρόταση να είναι κανείς δηλαδή περισσότερο γενναιόδος για να καλύψει και μικρότερες καταστροφές από όσες προβλέπονται, αποβαίνει πάρα πολύ δύσκολο να περάσει. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε δημιουργικά να είμαστε Ουδέτερη και δεν θέλουμε να ανεβάζουμε τις προσδοκίες ή να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή. Το θέμα ειναι κατά πόσον εγκρίνει το Συμβούλιο, το οποίο πάντοτε ήταν διστακτικό για η πρόταση η οποία θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες δαπάνες. Το σχέδιο κειμένου της κυρίας Σεσταράς περιέχει διάφορα στοιχεία. Δεν είμαι βέβαιος εάν όλα αυτά τα οποία αναφέρει το κείμενο θα εξυπηρετήσουν τον επιδιωκόμενο σκοπό, δηλαδή το να τροποποιήσουμε το Ταμείο, τη λειτουργία του. πάντων. Έχουμε αυτά τα, τα ευέλικτα κριτήρια, αλλά στο Ταμείο παλεύουμε με διάφορες προϋποθέσεις που προβλέπονται και που προσφέρονται για πολλαπλές ερμηνείες. Έχουμε τώρα έναν διορθωτικό συντελεστή όσον αφορά το κριτήριο της κοινωνικονομικής κατάστασης πέραν του ΑΕΠ. Οπότε, με όλα αυτά, κάτι θα διαδυσχερέσει τη λειτουργία του Ταμείου και η πρόταση του κοινωνικού μας κειμένου είναι ακριβώς να διευκολυνθεί η λειτουργία. Η πρόταση επίσης να είναι περιοχή αναφοράς οι περιφέρειες του, του, του ΝΑΤΣ 3 με προβληματίζει, δεν ξέρω. εντάξει, έχουμε ως σημείο αναφορά στο ΝΑΤΣ 2, αλλά αν έχουμε ε, και μικρότερες περιοχές και περιφέρειες στο ΝΑΤΣ 2 και αυτές θα είναι επιλέξιμες. Είτε είναι όμορες είτε όχι. Αυτές είναι περιοχές του ΝΑΤΣ 2. Αν τώρα επομένως βάλουμε για το ΝΑΤΣ 3 ως αναφορά, τότε περιορίζουμε την ε, κινητοποίηση, τη δράση του Ταμείου. Είπαμε ότι οι εξόχους από τις περιοχές είναι περιοχές του. Δύο και μόνο θα καλύπτονται. Είπαμε να τονίσουμε και την κάλυψη αυτών των περιοχών γιατί τα κριτήρια της κινητοποίησης είναι ευέλικτα. Κοινωνικο-οικονομικά. Τώρα προσθέτουμε ή προ, προτείνεται τέλο πάντων αυτό το κατόφλι κινητοποίηση που σχετίζεται με το ΑΕΠ. Δεν ξέρω πώς αυτό κολλάει στο ότι πρέπει να προσέξουμε ή να καλύψουμε καλύτερα τις εξόχους απογοήτες περιφέρειες. Είναι θέμα κατοφλίου ίσως. Επίσης, η να καλυψουμε καλυτερα τις από απογοητες περιφερειες ειναι θεμα κατοφλιου ισως επισης η αυξηση των προκαταβαλωμένων. Και αυτό σηκώνει συζήτηση. Θα μπορούσε να είναι θετικό. Όπως και η παράταση της σχετικής περίοδου από 12 στους 18 μήνες. Βέβαια, εάν παραταθεί αυτή η περίοδος εφαρμογής, αυτό σημαίνει ότι ακυρώνουμε αυτό το οποίο θέλουμε, γιατί εμείς θέλουμε να καταστεί ταχύτερη η παρέμβαση του Ταμείου, να πληρώνει πιο γρήγορα. Εάν πάμε στους 18, μας 15 εβδομάδες ας πούμε που προσθέτουμε, τότε αργεί η παρέμβαση του Ταμείου και δεν ξέρω επομένω εάν αυτό θα βοηθούσε, εάν συνάδει προς τις προθέσεις μας. Ξέρουμε ότι 10 εβδομάδες είναι σχετικά μικρό διάστημα, αλλά ανέκαθεν δεχόμαστε επιπλέον πληροφορίες ε, και είμαστε ευέλικτοι με αυτές τις προθεσμίες. Άρα καλύτερα να είμαστε ευέλικτοι με την προθεσμία παρά να ξεκινήσουμε προβλέποντας μια παρατεταμένη τέτοια περίοδο εφαρμογή και παρέμβαση. Τώρα, το Ταμείο Αλληλεγγύης. Όταν συγκροτήθηκε έγινε για να μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη. Επομένω, το, το, το, σημείο είναι τα κρατη τα κρατη και όχι οι περιφέρειες, ούτε καν οι ε, ούτε του καν διασυνοριακά. Επομένω, το Ταμείο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα κράτη-μέλη ε, για τι δυσκολίε που έχουν αντιμετωπίσουν μετά από κάποια καταστροφή, θεομηνία κλπ. Εάν τώρα προσθέσουμε και αυτή τη λειτουργία την διασυνοριακή, αυτό θα δυναμητήσει όλο το σύστημα, όλο το οικοδόμα και δεν ξέρω πώς θα υλοποιηθεί μια τέτοια πρόβλεψη. Τα κατόφλια σε σχέση με το κράτος μέλος κλπ. κλπ. Θα είναι τελείως καινούργιο χαρακτηριστικό. Που δεν συνάδει, δεν ταιριάζει με την αρχιτεκτονική που έχουμε κατά νου. Άλλο μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος, όχι παραπάνω. Καλά, καλά. Βάζω τελεία τότε εδώ και τώρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπράντα, θέλετε και εσείς το λόγο. Και κατόπιν θα κλείσει η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ στομή η πρώτη μου τοποθέτηση. να και είμαι εδώ. Πολλά θέματα ακούστηκαν για την ε, πρόληψη. Και συμφωνώ εδώ με την εισηγήτρια ότι τα μέτρα για την πρόληψη φυσικών καταστροφών έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Περισσότερη όμως ε, γραφειοκρατική ε, ταλαιπωρία, επιβάρυνση μπορεί να προκύψει από την στενή προθεσμία των 10 εβδομάδων. Μέσα σε 10 εβδομάδες μόνο από την ώρα που έχει έρθει όλη αυτή η καταστροφή πρέπει κανείς να έχει ολοκληρώσει όλη τη διαδικασία. Ε, νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει. Επιβαρύνει πολύ περισσότερο και βέβαια δεν βοηθάει και στο στόχο της πρόληψης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει η νομοθεσία καταρχάς να αναφέρεται ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία, ε, να καλυφθούμε από την οδηγία για τις ε, πλημμύρες και να δούμε τι είδους πληροφορίες χρειάζονται, απαιτούνται ως βασική κατάθεση, ως βάση για την κατάθεση μιας αιτήσεως και μετά να δούμε πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόληψη. Ευχαριστώ πολύ. Άννα. Εισηγήτρια, ευχαριστώ πολύ. Έτσι είναι. Η προτεραιότητα είναι η πρόληψη. Ακριβώς όπως ε, έλεγχε το αρτίκολο 4F το οποίο καταργήθηκε ε, πάνω σε αυτό έχει δίκιο ο κύριο Μπράντα από την Επιτροπή των Περιφερειών. Όταν κανεί θέλει να παρουσιάσει κάποιε πληροφορίε, θα πρέπει κανεί να, να, να περιγράψει ότι τι εννοούμε, τι θα πει, ε, τι θα πει πρόληψη. Ε, θα πρέπει πάντω όταν κάποιο ζητεί βοήθεια να το αιτιολογήσει. Δεν γίνεται γενικόλογα τέλο πάντων το αίτημα βοηθεία. Αλλά πρέπει κανεί να παράσχει τις λεπτομέρειες. Είπαμε γι' αυτό το 1% για τις περιφερειακές καταστροφές. Και αυτό αφορά το περιφερειακό ΑΕΠ. Και επίσης αυτό συνδυάζεται με κοινωνικονομικά κριτήρια, ούτως ώστε να μην έχουμε κάποιους που θα υποστούν καταστροφή και δεν θα καλυφθούν. Έχουμε το 1,5%, το 1% προτείνουν μεν και ιδέα, αυτό θα περάσει από τον τριγωνικό διάλογο. Όσο νωρίτερα συμφωνήσουμε, τόσο καλύτερα. Όσον αφορά τώρα το ΝΑΤΣ 3, είπαμε, όπως και η Επιτροπή των Περιφερειών, να μπορούμε να καλύψουμε και αυτό τον κόσμο, όπως και στο ΝΑΤΣ 2. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις ε, παραμεθόρες περιοχές ή τις ε, διασυνοριακές περιφέρειες. Όλα αυτά χωρίς να υπονομεύσουμε το Ταμείο. Οι διασυνορικές περιοχές πάντοτε ζητούν το να καλυφθούν και είπαμε γι' αυτό το 1% να καλύπτει και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. 10 με 15 εβδομάδες και 18 αντί για 12 μήνες όσον αφορά την εφαρμογή για την, την τη της ενίσχυσης. Όχι, εμείς θέλουμε να δώσουμε χρόνο στο κράτος μέλος για να κάνει τις κατάλληλες τεχνικές μελέτες, για τις ζημίες, για το κόστος το οποίο απαιτείται. Βεβαίω και χρειάζεται η άμεση βοήθεια. Αλλά είπαμε να δώσουμε αυτό το περιθώριο των 5 εβδομάδων. Ε, Θέλουμε έτσι να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο στην περιφέρεια αλλά και στα θύματα. Θα πρέπει να ε, δούμε ε, έχουμε την ακρόαση, έχουμε την τροπολογία της, ε, την τροπολογία της 6 Ιανουαρίου και άρα θα πρέπει να γίνουν οι τριμερείς αντίσεις με συμβουλευτική Κομισιόν και να δούμε το Μάρτιο πώς θα γίνει να περάσει αυτό το κείμενο. Δεν είδα Μαριτερές που είχες δει στο λόγο. Παρακαλώ Μαριτερές να μιλήσεις μόνο για ένα λεπτό, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τη Ρόζα και να υποστηρίξω και ε, τις προτάσεις της. Ε, η αλληλεγγύη είναι μία από τις ε, θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην το ξεχνάμε και όπως και ο κύριος Μπράντερ νομίζω πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, είναι βασική μέρη όλων. Θέλω να πω στην, στον πρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το θέμα δεν είναι η γενοδορία, είναι ακριβώ η αλληλεγγύη. Ο τώρα των φυσικών καταστροφών ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπερβάλλουμε, δεν έχουμε, και, έχουμε περιορισμένους πόρους. Προσυπογράφω ε, mm. την πρόταση ε, τα τεχνικά κριτήρια να ε, επισέρχονται στην επιλεξιμότητα. Τώρα για τις κλιματικές αλλαγές, ε, το να το συνδέσουμε με τις κλιματικές αλλαγές είναι λίγο επικίνδυνο. Πώς θα συνδέσουμε τον ορισμό με τις κλιματικές αλλαγές για να χαρακτηριστεί κάτι ως φυσική καταστροφή. Αφήστε που οι ασφαλιστικές εταιρείες ε, μέχρι να συμφωνήσουν για την ε, επανόρθωση των ζημιών χρειάζονται χρόνια ολόκληρα. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια έγκαιρη επέμβαση. Ε, τελικά θα ε, περικοπεί ο προπολογισμό στο ίμιση και θα είναι πολύ περιορισμένη η επιλεξιμότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι, αλλά ξαναλέω ότι είναι προτεραιότητα για μας η αλληλεγγύη. Το Συμβούλιο πρότεινε περικοπή γιατί δεν απορροφούνται τα κονδύλια. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι εύκολη η πρόσβαση. Ας κατεβάσουμε τα όρια τότε. Ε, κοντά στη Λούρδη ε, στη, και στην νοτιδυτική Γαλλία γενικά θα μπορούσαν να είχαν υποφεληθεί από το Ταμείο αν ήταν διαφορετικά τα όρια. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. 7 πρώτου 12 είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες. Λοιπόν, μας έχει μείνει λίγο λίγος χρόνος για την έκθεση της κυρίας Αβίσα Τόμας. Ε, ε, είμαστε στο στάδιο ε, της εξέτασης των συμβαστικών τροπολογιών και πρόκειται για την 7η και 8η έκθεση συνοχής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Πιστεύω ότι όλοι είσαστε υπατμών να γυρίσετε, να γιορτάσετε στις πατρίδες σας η έκθεση αφορά την 7η και 8η έκθεση πρόοδου για την πολιτική της συνοχής. Και βέβαια και την υλοποίηση των προγραμμάτων 2012-2013. Οι τροπολογίες για μένα μετά το πρώτο σχέδιο που συνέχισα να επεξεργάζομαι το κείμενο ε, έχουν καταρχάς προέρθει από μένα, οι, περισσό, οι μισές τουλάχιστον, έχω κάνει κάποιες διευκρινήσεις από πράγματα που είδα. Άλλωστε τα είχα επισημάνει και κατά την ε, παρουσίαση της έκθεσης. Ο κύριος Μιθ έχει κάνει κάποιες προτάσεις, αλλά δεν βλέπω τώρα εδώ. Ο κύριος Ντόιτς επίσης φαίνεται να φύγε πριν αρχίσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. κύριος Βλάσακ επίσης έχει κάνει ε, τροπολογίες αλλά δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες. Θα έχετε όλα γραπτός. Πάντως εγώ τις κοίταξα, τις μελέτησα, τις τροπολογίες του κύριου Βλάσακ και μπορώ να εκφράσω ήδη τις ευχαριστίες μου. Ξεκινώ με αυτό λοιπόν. δεν είμαι κατά των τροπολογιών. Μπορώ να τις υποστηρίξω. Αλλά δεν θέλω να χάσει και τη συνοχή και τη συντομία ε, το κείμενο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να καταθέσω ε, για τις αρχές Ιανουαρίου κάποιες ε, τροπολογίες στις οποίες θα ε, συλλέξω τις τροπολογίες για να δουλέψουμε σε ένα κοινό κείμενο. Ο κύριο Ντόιτ δεν είναι εδώ, ο Γιέντς όμω είναι εδώ. Ο Γιέντς είναι στον εκ σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Έχω καταθέσει πολύ έρευνε τροπολογίες, 8-9, αν θυμάμαι καλά. Ε, αυτές οι εκθέσεις που επί ιστορικών δεδομένων ε, δεν είναι κάτι που πρέπει να αγνοούμε, γιατί από την ιστορία μαθαίνει κανείς για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικέ πληροφορίε που υπάρχουν μέσα σε εκθέσει συνοχή. Όταν έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε τι έχουμε κάνει τα τελευταία 7 χρόνια, ε, για να σχεδιάσουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο μέχρι το 2020, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε τη δράση μας. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όλες ε, τις τροπολογίες. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω μόνο κάτι που τονίζετε και εσείς στην έκθεση, ότι υπάρχει μια κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που δεν λαμβάνουμε δεόντως ε, υπόψη και αυτό θα έχει αξιανόμενη σημασία και για το μέλλον. Ο Πάκανίναν έχει καταθέσει πολύ καλές τροπολογίες. Εάν η συγγήτρια τη λάβει υπόψη και λάβει υπόψη και τι δικέ μου τροπολογίε, θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ, Ότσο Βλάσεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ε, συμφωνώ πλήρω με την συγγήτρια. Είτε πρόκειται η θετική είτε για αρνητική αξιολόγηση, ε, η αξιολόγηση στην οποία θα καταλήξουμε απαιτεί πολύ αξιόπιστες στατιστικές, στατιστικά στοιχεία. Πρώτον. Δεύτερον, το reporting, η υποβολή των εκθέσεων θα μπορούσε να καταστεί υποχρεωτική. Και έτσι καλό θα να υπάρξει μια διατύπωση η οποία να καλύπτει αυτό το θέμα χωρίς όμως να, ε, να επεκτείνει πολύ το πεδίο του ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Κύριο Αλφονσί. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση διότι υπογραμμίζει όλα τα μειονεκτήματα της πολιτικής συνοχής, την ανεπάρκεια των κονδυλίων, την όχι πολύ καθαρή ματιά στις ανάγκες. Σε αυτό λοιπόν συμφωνούμε. Απλώς μας προβληματίζει ως ομάδα αυτή η αναφορά σε μια κατακόρυφη ε, μέθοδο. Ξέρετε ότι εμείς προτείνουμε πάντα τις εγκάρσεις μεθόδους, δηλαδή στην κατάρτιση των προγραμμάτων ε, να μην χρειάζεται να περνάμε από τις κρατικές υπηρεσίες αλλά από τις περιφερειακές. Φυσικά ένας κανόνας μπορεί πάντα να έχει εξαιρέσει, αλλά όταν οργανώνεται ένας ε, κανόνας ε, δεν πρέπει να πολλαπλασιάζονται οι εξαιρέσει. Αυτό λοιπόν το κομμάτι νομίζω ότι σωστά πρέπει να καταργηθεί. Αυτό εκ μέρους μας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητεί κανείς άλλο το λόγο. Ο Τζον Βόλφ όμως νομίζω ήταν ε, εδώ εκ μέρους της Επιτροπής για να σχολιάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ με την εισηγήτρια και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για τις τροπολογίε Η στρατηγική έκθεση είναι μέρος του πακέτου και έξω και η πολυπλοκότητα της εκμόνωσης μιας τέτοιας έκθεσης ε, αποτελεί με ένα στιγμιότυπο, μια έκθεση πρόοδου ε, ως προς την εφαρμογή ε, της πολιτικής συνοχής των 347 δις. Ε, βλέπουμε λοιπόν το τι έχει επενδυθεί, τη ροή των επενδύσεων για την πρόληψη των κινδύνων, για την έρευνα, όπως είπε ο συνάδελφος, για την αγορά εργασίας, για την κοινωνική ένταξη και το καθεξής ε, και δικαίω η έκθεση αναφέρεται σε στοιχεία κλειδιά που καλύπτονται και στη στρατηγική έκθεση αλλά και στην 7η και 8η έκθεση προόδου. Ε, συζητήσαμε το, το αρχικό σχέδιο της έκθεσης ε, και βλέπουμε ότι στην 7η και 8η έκθεση εξετάζουμε σε περιφερειακό επίπεδο τις, ε, κοινωνικο-οικονομικές τάσεις χρησιμοποιώντας δεδομένα της Eurostat ε, για αυτές τις τάσεις. εξετάζουμε και τον τρόπο συλλογής αυτών των δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο. Καλά κάνετε και τονίστε ότι επιδέχεται το σύστημα περαιτέρω βελτίωσης και έχουμε ήδη αναλάβει δέσμευση περί αυτού. Τώρα για τα θέματα που σας αποσχολούν απασχολούν. Βλέπουμε και εξετάζουμε τις επιπτώσεις κοινωνικο-οικονομικής κρίσης. Στην 8η έκθεση βλέπετε ότι η κρίση είχε πολύ διαφορετική και επιπτώσεις ως προς το βαθμό σοβαρότητας ανάλογα ε, με τις περιοχές ε, και τα κράτη-μέλη. Ε, σωστά κάνετε και εξετάζετε τις επιπτώσεις για τη μελλοντική πολιτική συνοχή. τονίζετε τη σημασία της υποδομής. Άλλοι πάλι ασχολείται με την υποστήριξη των επιχειρήσεων, την καινοτομία και την έρευνα και σίγουρα είναι ε, ευπρόσδεκτη η υποστήριξή σας για την ευφυή εξειδίκευση ε, και ε, των καλύτερων περιφερειακών πολιτικών εξειδίκευσης. Επίσης, η σημασία των συνεργατικών σχέσεων, δηλαδή η εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο σχεδιασμό των μελλοντικών πολιτικών έχει ιδιαίτερη σημασία και ο κώδικας ιδιωτολογίας για τέτοιες εταιρικές σχέσεις είναι κάτι που συντάσσουμε αυτή αυτή τη στιγμή ε, ακολουθούμε δηλαδή την ίδια κατεύθυνση όπως και εσείς στην έκθεση. Επίσης ε, θα μπορούσαμε να πούμε ε, όπως και εσείς το λέτε ότι ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα για την εποπτεία ε, όντως με κάθε στιγμή ότι έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα, μια φωτογραφία καλύτερης ανάλυσης. συνεργαζόμαστε με τις διαχειριστικές αρχές και βλέπουμε ότι με το ΕΤΠΑ έχουν δημιουργηθεί 600 200.000 θέσει απασχόληση, ε, τουλάχιστον ε, Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, θέλουμε να αυξηθεί η διαφάνεια. Ξέρουμε ότι συνεπάγεται μεγαλύτερο άκθο, αλλά ε, χρειαζόμαστε διαφάνεια για να αντλήσουμε τα διδάγματα ω προς τη μελλοντική πολιτική και να χρησιμοποιούμε ορθότερα τα διδάγματα του παρελθόντο. Ευχαριστούμε πρώτα, ευχαριστούμε και την εισηγήτρια. Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Θέλει η εισηγήτρια μήπως να απαντήσει σε αυτά τα σχόλια του εκπροσώπου τη Επιτροπή. κομμεντάρι, πώ ja ja τον ja ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Βλέπω ότι είναι πολύ θετικά και ενθαρρυντικά όλα τα σχόλια. Η ΔΕ Επιτροπή συνόψε πολύ αποτελεσματικά την ουσία των τροπολογιών. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Θέλω απλώς να πω και πάλι στους αδέλφους ότι θα επανέλθω με τροπολογίες το ταχύτερο δυνατό και ελπίζω να μην υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Για τις 22 σκοπεύουμε στην προσοχή μας συνεδρίαση. Να κάνουμε την έγκριση, την ψηφοφορία. Περνάω τώρα στους συντονιστές, έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι έχει κλείσει τώρα το θέμα. Έχουμε το απόγευμα μόνο τη συνεδρίαση. Σημαντική συνεταιρία στο απόγευμα. Παρακαλώ να είστε όλοι παρόντες. Προς το παρόν συντονιστές.